Uh, Κυρίες αλλά και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε αργήσει και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με μεγάλη χαρά δίνω χαιρετίζω τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τα θέματα εσωτερικής αγοράς και έχουν να μας ε, παρουσιάσουν μια σειρά από θέματα όπου έχουμε μεγάλη εμπλοκή και εμείς ως Επιτροπή ΙΜΚΟ διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς, αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς και το μέλλον του λύσετου του Solvit δηλαδή. Με μεγάλη χαρά λοιπόν τους ε, χαιρετίζουμε. Όπως ξέρετε συνεργαζόμαστε ιδιαίτερα <clears throat> για να προχωρήσουμε στα θέματα της ε, εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τα χείλη της εκπροσώπου της Κομισιόν ποιες είναι οι νέες τους ιδέες στα θέματα αυτά. Θα δώσω λοιπόν στην Κομισιόν το λόγο για να κάνει μια παρουσίαση προς εμάς εγώ θα την κάνω στα κάτω εδώ για να βλέπω καλύτερα, γιατί αυτή τη στιγμή σας εμποδίζω τη θέα στην οθόνη. Και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Μόλις τελειώσετε, σας δίνω λοιπόν το λόγο και σας αδειάζω τη γωνιά για να μπορέσετε να κάνετε την παρουσίασή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι γνώμων που μου δίνετε τέτοια ευκαιρία να προσέλθω διότι αυτά είναι σαν διαφήμιση για την έκθεσή μας, για το check-up. Θέλω να σας εξηγήσω πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εσείς εδώ στην Επιτροπή σας μερικές φορές παίρνατε διάφορες εκθέσεις μας για συγκεκριμένες πτυχές της εσωτερικής αγοράς όπως το scoreboard ή εκθέσεις IMI. I've become increasingly aware that... Και τελικά φάνηκε ότι είναι πολλές αυτές, πολλές και υπερβολικά πολλά στοιχεία και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να βάλουμε σε μια σωστή προοπτική το θέμα της governance της εσωτερικής αγοράς. Δεν είναι η πρώτη μας έκθεση, είναι η μηδενετική. Είναι πείραμα. Εγώ λοιπόν με την ομάδα μου εδώ και δίπλα μου έχω και την Μάριον είπαμε ας δούμε τα πράγματα πιο ολιστικά τον Gestalt να δούμε δηλαδή το σύνολο του κύκλου ζωής της governance από τις ιδέες μέσω της νομοθεσίας μέχρι και την πραγματοποίησή της. Πραγματοποιείται, εφαρμόζεται σωστά, μήπως χρειάζονται αλλαγές. Όλον αυτόν τον κύκλο της governance θελήσαμε να δούμε. Να δούμε πώς γίνεται η μεταφορά της νομοθεσίας, πώς πληροφορούνται οι επιχειρήσεις και οι λαοί πώς οι δημόσιες αρχές συνεννοούνται καλύτερα, πώς λύνουν προβλήματα ενιαίας αγοράς, πώς αξιολογούν και ε, κρατάνε στα αρχεία τους ε, τις πληροφορίες και πώς χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για τη λήψη νέων αποφάσεων. Σε αυτόν τον κύκλο λοιπόν βλέπετε ότι, ότι σε διάφορες φάσεις του κύκλου γράφουμε εκθέσεις και πληροφορούμε. Βλέ, παρατηρούμε, εποπτεύουμε τη μεταφορά της νομοθεσίας. Έχουμε τα σημεία όπως το Hugo και αν τυχόν συμβεί, επισυμβεί κανένα πρόβλημα έχουμε το σύστημα λίστο, it. Και αν τα πράγματα πάνε ακόμη χειρότερα, έχουμε και το σύστημα επίλυσης διαφαρών με το δικαστήριο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ερχόμαστε και σε εσά σας πληροφορούμε, γιατί έχουμε τα στοιχεία, τα στοιχεία. Διότι έχετε πει και εσείς ότι θέλετε η λήψη αποφάσεων να βασίζεται σε στοιχεία. Έτσι έχουμε ένα σωστό και ολοκληρωμένο προϊόν. Αποφασίσαμε λοιπόν να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις εκθέσεις και αξιολογήσεις και δημιουργήσαμε μία fitness check. Ένα, μία δοκιμή ευρωστίας. Για κοιτάξτε αυτή τη δοκιμή ευρωστίας. Όπου βλέπετε πράσινο να χαίρεστε. Όπου είναι κίτρινο κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και τα κόκκινα είναι πρόβλημα. Η όλη λοιπόν διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς φαίνεται στα κόκκινα. Από εκεί βλέπετε ότι έχουμε πολλά προβλήματα γιατί έχουμε πολλά κόκκινα. Μόνο μία χώρα μέλος είναι κατά πράσινη, η Εσθονία. Και σε σχετικά καλή κατάσταση η Λετωνία, η Σουηδία, η Δανία και η Λιθουανία. Πρέπει όμως να σας πω ότι παντού αλλού χρειάζονται βελτιώσεις. Είναι λοιπόν πολύ μέτρια η ιατρική αναφορά. Για να δούμε τώρα για την μεταφορά της κοινοτικής ναμαθεσίας. Εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει χειροτερέψει σε σύγκριση με πέρυσι. Αλλά ακόμα μένουν και πολλές οδηγίες να μεταφερθούν. 48% των χωρών μελών είναι στο κόκκινο. Και μετά για τις παραβιάσεις έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά ο αριθμός τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο 37% των χωρών μελών είναι πάλι στο κόκκινο. Τώρα η διάρκεια των παραβιάσεων είναι μεγαλύτερη. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Και για το Your Europe που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για όλα τα υπήρξε κάποια πρόοδος μεν 37% δηλαδή των πληροφοριών που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη είναι σωστά, σωστές πληροφορίες και μόνο το 19% είναι κακής ποιότητος ή λύπη τελείως. Σχεδόν τα μισά κράτη-μέλη όμως πρέπει να μας δίνουν σαφέστερες πληροφορίες. Επίσης για το Your Europe Έχουμε εκείνο το σύστημα ελεύθερης ή δωρεάν διαβούλευσης. Αυτό πάει καλά. 15.000 περιπτώσεις έχουν τύχη διαβούλευσης. 15.000 ερωτήματα τέθηκαν. Αλλά ακόμα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Πάντοτε ακούγονται παράπονα για την εθνική και ενωσιακή διοίκηση, γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρξει μεγάλη βελτίωση. Για τα single points of contact ή points of single contact, εδώ είναι θέμα εφαρμογής της οδηγίας των υπηρεσιών. Και λέει, βλέπουμε εδώ ότι μόνο 26% ένα τέταρτο είναι εντάξει. 22% δεν λειτουργούν σχεδόν καθόλου και τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Άρα πρέπει ακόμα να χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά και για τα single points of contact. Όποτε πρόκειται για πρόβλημα μετακίνησης, ε, πρόβλημα από μια χώρα στην άλλη, θα περίμενε κανείς περισσότερα μεταφρασμένα κείμενα, αλλά δυστυχώς το 70% των επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν τίποτε για όλα αυτά. Και τώρα το IMI. Εδώ 40% χρησιμοποιούν το σύστημα πολύ καλά για τα επαγγελματικά προσόντα και λοιπά. πάνω από τις μισά ερωτήματα απαντιούνται μέσα σε δύο εβδομάδες και υπάρχει πρόοδος για τον κανονισμό του IMI. Ό,τι αφορά βέβαια την εφαρμογή της οδηγίας των υπηρεσιών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και μερικές χώρες μέλη απαντούν, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να απαντήσουν. Τώρα για το λίστο το Solvit, εδώ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η δοκιμή ευρωστίας έδειξε ότι σχεδόν 70% πάνε καλά, 27% χρειάζονται βελτίωση και 5% έχουν πρόβλημα κυρίως λόγω ανεπαρκούς προσωπικού αριθμού. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι από αυτό το πρόβλημα του προσωπικού εξαρτάται σχεδόν το σύνολο της επιτυχίας του Solvit. Ακόμη και αν τα πράγματα είναι καλά λοιπόν υπάρχουν εδώ λόγοι ανησυχίας. προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια δεύτερη γενιά Solvit. Υπάρχει μια στρατηγική που καταστρώθηκε με 10 βήματα βελτίωσης. Για το IMI υπάρχουν νέα εργαλεία πληροφορικής που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο και θα διατυπώσουμε προτάσεις για το Solvit στα τέλη του έτους. Αυτά είχα να σας πω. Ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν όλα αυτά. Γιατί έπρεπε να συμφωνήσουν οι συντάκτες όλων των εκθέσεων που είχαμε ποτέ συντάξει. Τελικά όμως φάνηκε ότι στην Κομισιόν είπαν όλοι και εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε στην έκθεση αυτή του χρόνου λοιπόν που θα αναλύσουμε τις προοπτικές των επιχειρήσεων θα προσπαθήσουμε όπως κάθε φορά να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αλλά με τρόπο ευνόητο, εύληπτο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τα μάλα. <clears throat> Νομίζω ότι έχετε ανταποκριθεί πλήρως στις ανησυχίες των βουλευτών για το θέμα της παροχής ε, πληροφοριών και εκθέσεων και την ε, υπερφόρτωση κατά κάποιο τρόπο με πληροφορίες που έχουμε μερικές φορές. Εγώ θα επανέλθω στον τόπο μου, αλλά προηγουμένως Έχουμε κάποια ερωτήματα. Βλέπω ο κύριος Σουάπ και η κυρία Γκέπχαρτ να είναι εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να χαιρετήσω την κυρία Κολίν Λάγκεν, η οποία αντικαθιστά τον κύριο Λέσνερ. Είναι, ήταν πρώην δήμαρχος μιας σημαντικής πόλης στη Ρινανία και εκτός από την εμπειρία της μπορεί να μοιραστεί μαζί μας και τα θαυμάσια κρασιά της περιοχής της. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σχόλια. Κύριε Σουάμπ, θέλετε να πείτε κάτι. Και τώρα που έφυγε και η οθόνη μπορούμε να επανέλθουμε στις θέσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ντέιλι, σήμερα το πρωί με ένα αξιοσημείωτο τρόπο κατέδειξε ποιε είναι οι αδυναμίες της υποδομής της ενιαίας αγοράς και γι' αυτό της είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Πιστεύω ότι αυτό είναι και ο στόχος μας εδώ να μπορέσουμε να βρούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις αδυναμίες στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ ότι το θέμα της ε, ευκυβερνησίας της ε, νέας αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχε τονίσει και ο καθηγητής Μόντι όταν ήταν επίτροπος ότι είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την ενιαία αγορά. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όμως είναι να δούμε ποια είναι τα είδη δικτών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γίνει πιο απτή η αναζήτηση της ευκυβερνησίας στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Η ομάδα του ΕΛΚ έχει δημιουργήσει το φόρουμ της ενίας αγοράς όπου μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Θέλω λοιπόν να θέσω αυτό το ερώτημα στην κυρία Ντέιλι. Τι ρόλο παίζει για σας το Single Market Forum σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, η δοκιμασία ευρωστίας που την έχετε παρουσιάσει σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, αυτό είναι πολύ ωραίο και χρωματιστό. Κάθε χρόνο φυσικά είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα θέλαμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα από ό,τι μας δίνει αυτό το γράφημα, Ποιε είναι οι πραγματικές διαρθρωτικές αδυναμίες που υποκρύπτονται πίσω από τα κόκκινα χρώματα και επίσης να δούμε κατά πόσο το σύστημα Solvit έχει πραγματικά λειτουργήσει σε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως και στις χώρες που υπάρχει πράσινο υπάρχουν σημεία που πρέπει να χρωματιστούν κίτρινα ή κόκκινα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της τελευταίες συνεδριάσεις του έχει τονίσει ότι το κύριο μέτρο το κύριο μέσο μάλλον για την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι η εσωτερική αγορά και πρέπει να την ενισχύσουμε περισσότερο. Επομένω, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη την ευθύνη που έχουν για την ευρωστία και την ενίσχυση τη εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποιε είναι οι καταστάσει σε σχέση με την στελέχωση με προσωπικό των υπηρεσιών του Σόλβιτ σε ορισμένα κράτη-μέλη, που υπολείπονται. Κύριε Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντέλη για τι πληροφορίε που μα έδωσε. Ήθελα να κάνω μια παράκληση προς την κυρία Ντέιλι να μας στείλετε και τις διαφάνειές σας, τις έχουμε μονάχα σε μαυρό άσπρο και χάνουμε τη χρωματική παλέτα που περιείχε το, η παρουσίασή σας. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε λοιπόν και τις διαφάνειές σας. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία έχουν απασχολήσει την Επιτροπή μας και φυσικά όλο το Κοινοβούλιο είναι το θέμα αυτό της ευκυβερνησίας. Μας ενδιαφέρει εφόσον έχουμε καταβάλει τόσο καλή προσπάθεια για τα θέματα αυτά να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια σωστή διοίκηση και διαχείριση των θεμάτων αυτών. Υπάρχουν μερικά σημεία ιδιαίτερα που αφορούν το, την μοναπευθυντική θηρίδα, το, το μοναδικό σημείο στο οποίο πρέπει να απευθύνεται κανείς θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας, για τους βουλευτές μας, αν θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποια είναι τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στο κόκκινο. Μας ενδιαφέρει κάπως λιγότερο αυτό που έχει να κάνει με τις χώρες που είναι στο πράσινο. Αυτές λειτουργούν καλά, αλλά εκεί που υπάρχουν προβλήματα, οι χώρες που βρίσκονται στο κόκκινο, <clears throat> θα θέλαμε να ξέρουμε σε ποια σημεία παρουσιάζονται προβλήματα και πώς προκύπτουν. Είναι θέματα ε, στελέχωσης με προσωπικό, είναι θέματα υποδομών, είναι θέματα γλωσσικά, είναι θέματα μη δημιουργίας ε, ιστοσελίδων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον πολίτη και τον καταναλωτή. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν κάποια περισσότερα στοιχεία για το γιατί δεν λειτουργεί η κατάσταση σε ορισμένε χώρες. Στη δική μου περιοχή, στην Βάδη Βιτεμβέργη, είναι πάρα πολλέ αυτέ οι υπηρεσίε ίσω και μπορεί και αυτό να είναι ένα πρόβλημα. Ο πολίτη δεν ξέρει ακριβώ πού πρέπει να απευθυνθεί. <clears throat> ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να αντιμετωπίσω είναι το Solvit και η σύνδεσή του με το σύστημα IMI. Είπατε ότι το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να έχουμε τα εργαλεία αυτά στη διάθεσή μας. Τα ήλπιζα και εγώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί για το σύστημα IMI συζητάμε εδώ και χρόνια. Κάθε χρόνο έρχεται κάποιο από την Κομισιόν, ο οποίο μας παρουσιάζει την πρόοδο και λέει του χρόνου, μα σίγουρα του χρόνου θα δουλέψει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. <clears throat> και θα είναι λειτουργικό και θα μας ικανοποιήσει όλους τους τομείς που μας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα όμως να ξέρω από εσά μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από τόσες δυσκολίες που αντιμετώπισε το IMI για να εφαρμοστεί, θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινά αν είμαστε πραγματικά σε σημείο που να είναι έτοιμο αυτό το σύστημα ή αν ακόμα παραμένουν κάποια προβλήματα. Θέλετε να θέσετε κάποια ερωτήματα και οι υπόλοιποι από μένα, αν μπορώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Όλα αυτά είναι πολυθετικές εξελίξεις που παρουσιάσατε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για περαιτέρω πρόοδο για μένα ένα τμήμα του προβλήματος στα θέματα της εσωτερικής αγοράς είναι και το να μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε τους δείκτες σε σχέση με την σημασία τους. Όταν μιλάμε για το ποσοστό μεταγραφής των νομοθετημάτων, αυτό είναι πολύ περισσότερο για την ε, ενιαία αγορά αν ένα σημαντικό νομοθέτημα έχει μεταγραφεί με λαθασμένο τρόπο και λιγότερο πρόβλημα αν είναι κάποιο τεχνικό θέμα. Μπορεί να δείχνουν λοιπόν στατιστικές το επίπεδο μεταγραφής, αλλά δεν είναι σαφές τι έχει γίνει με τα μεγάλα, τα σημαντικά νομοθετήματα για την ενιαία αγορά. Καταλαβαίνω είναι πολύπλοκο πρόβλημα, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό. Επίσης, ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αγορές και τα σημεία, ε, τα μονοαπευθυντικά σημεία, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να βελτιστοποιήσουμε τι δυνατότητε τη αγορά. Επομένω, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στι χώρε που έχουν μεγάλο δυναμικό αγορά, ώστε αυτά τα μονοπευθυντικά σημεία επαφή να λειτουργούν καλύτερα. Μία άλλη παρατήρηση. Είπατε στην παρουσίασή σα, κυρία Ντέιλι, ότι αυτά τα σημεία μονοπευθυντική επαφή ήταν σχετικά άγνωστα μέσα στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που έχουμε τονίσει έναντι τη Κομισιόν <clears throat> και η έκθεση της κυρίας Κιεπχάρτ για την εφαρμογή της ε, εσωτερικής αγοράς ήταν ιδιαίτερα επικριτική γιατί τα κράτη-μέλη δεν δίνουν στις επιχειρήσεις αυτή τη νέα δυνατότητα να έχουν κάποια καλύτερη πρόσβαση στην ενιαία αγορά με την μεταγραφή της ε, οδηγίας <clears throat> για την παροχή υπηρεσιών. Επίσης για το βαθμολόγιο της εσωτερικής αγοράς που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό είχαμε κάποιες προηγούμενες μορφές <clears throat> του βαθμολογίου όπου υπήρχαν και πληροφορίες σε σχέση με έρευνες που έλεγαν για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Για μας είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό <clears throat> σημείο καταμέτρησης πρόοδου για τα κράτη-μέλη, το αν υπάρχει πραγματικά πρόσβαση στην πληροφορία. Αν είχαμε μια επιχείρηση και λέγαμε τώρα στέλνουμε, φέρουμε στην αγορά ένα νέο προϊόν που είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες. Φτιάνουμε νέες ιστοσελίδες, αλλά δεν κάνουμε τίποτα σε επίπεδο marketing. Τότε χάνουμε τις επενδύσεις μας. Είναι σαν ελληνικά ομόλογα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι πολίτες στα κράτη-μέλη θέλουν όταν κάνουν επενδύσεις, όταν έχουν γίνει προσπάθειες για το Solvit, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις τεχνικές. Αν λοιπόν οι πολίτες και οι πελάτες δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά, δεν προχωρούμε. Γι' αυτό τονίζω την ανάγκη του να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για τους πολίτες. Όπως είπατε και εσείς, ήταν απογοητευτικό το επίπεδο ε, χρήσης του συστήματος IMI σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις ή άλλες διοικητικές διαδικασίες. Και αυτό μου δείχνει εμένα <clears throat> ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ευκαιρίες που δίνει η οδηγία για τις <clears throat> υπηρεσίες. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από κάποιες ε, περιορισμένες και κάπως μεροληπτικές στατιστικές καταμετρήσεις. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Οι άλλοι συνάδελφοι θα θέλαν να πούνε τώρα κάτι. Εάν όχι, σας δίνουμε και πάλι το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω για τους δείκτες, τι ακριβώς θα εννοούμε με αυτούς, τι ακριβώς θα καταμετρούν ως προς την αγορά. Αυτό που παρατηρήσατε πραγματικά λοιπόν εδώ είναι εύστοχο. Νομίζω υπάρχει ένας κίνδυνος παρόλα αυτά. Εάν επικεντρωθούμε μόνο στις παραβιάσεις, την μεταφορά και την υλοποίηση, ακολουθούμε δύο διαφορετικούς νομικούς δρόμους και μπορεί στη διαδικασία να ξεχάσουμε την οικονομική συνιστόσα. Πρέπει να εντοπίσουμε μια σωστή ισορροπία λοιπόν εδώ. Να έχουμε δείκτες που να καταμετρούν αυτά που μας ενδιαφέρουν σε σχέση με τις επιχειρήσεις, την κοινότητα των επιχειρήσεων και εταιριών. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ήδη προβλέψει για τη μελλοντική έκθεση. Επίσης, κατά καιρό συμπεριλαμβάνουμε κεφάλαια για θέματα όπως τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου, πώς αντιλαμβάνονται την ενιαία αγορά οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και ούτω καθεξής. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι το να δούμε τα προβλήματα που υποκρύπτονται, αυτό που αναφέρατε και στο πρώτο σας ερώτημα κύριε Σβάμπ, είναι να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αυτό αναζητούμε. Αυτό που κάναμε πέρσι, όταν καταρτήσαμε τον κατάλογο με τα 20 πρώτα προβλήματα, το top 20, είδαμε ότι αυτά που περισσότερο εκνευρίζουν τους ανθρώπους ε, στις, στην Ευρώπη, δεν είναι αυτά που τα, τα συζητούμε συνήθως στους διαλόγους που οργανώνουμε. Άρα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει οπωσδήποτε να τα συζητήσουμε στο μέλλον. Δεν ανέφερα καθόλου το φόρουμ, γιατί το θεώρησα περιττό, αλλά πραγματικά το φόρουμ ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, διότι είδαμε διαφορετικά επίπεδα ταυτόχρονα το πολιτικό, το διοικητικό και το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να υποτιμήσω το έργο μας βέβαια, αλλά υπάρχει πραγματικότητα. Δηλαδή, το τι στην καθημερινότητά τους αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πρόβλημα με την ενιαία αγορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι σαν ε, να μας ε, κρούει, να μας κρούει κάποιος στον κόδωνα του κινδύνου μια φορά το χρόνο για να δούμε την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, και φέτος, κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο, θα έχουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γίνεται με την ενιαία αγορά σε όλη την Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε με την Ολομέλεια εδώ στο Εμικύκλιο, αλλά ελπίζουμε ότι και οι βουλευτές θα συναντηθούν οι επίτροποι θα σκύψουν πάνω από το θέμα, οι εθνικοί βουλευτές και ιδίω τα κράτη-μέλη ότι θα συζητήσουν θέματα της ενιαίας αγοράς. Ως προς το IMI, λειτουργεί. Λειτουργεί και μάλιστα πολύ καλά. Εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία για το IMI, λειτουργεί σε πολλούς τομείς αποτελεσματικά το πιλωτικό πρόγραμμα για τα επαγγελματικά προσφαντά συγγνώμη για τη μετάθεση εργαζομένων, ήταν αυτό που μελετήθηκε και είδαμε ότι η... πολύ γρήγορα συλλέξαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μετάθεση εργαζομένων, την απόσπαση εργαζομένων στο IMI. Εάν σκεφτούμε ότι λειτουργεί σαν σιδηρόδρομος, σαν σιδηροδρομικό δίκτυο το IMI, κάποια από τα τρένα που θα ξεκινήσουν και θα λειτουργήσουν σε αυτό το δίκτυο θα αφορούν την απόσπαση εργαζομένων, κάποια τα επαγγελματικά προσόντα, αλλά Ουσιαστικά το σιδηροδρομικό δίκτυο αρχικά ε, καταρτίστηκε για τον οδηγία των υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να το αντιλαμβάνονται και δημόσιε αρχέ, πράγμα που δεν κάνουν ακόμη. Πρέπει να υπάρξει απαραίτητη διαφήμιση και προβολή για να καταλάβουν ότι αυτό είναι ο ευκολότερο τρόπο να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο. Κάτι που ίσω να μα έχει διαφύγει ω τώρα και είναι μια πραγματική πρόκληση, ο πρόεδρο εδώ το εντόπισε, είναι να καταλάβουμε την ε, σημασία των όσων κάνουμε σε όρους αγοράς. Αυτό μας απασχολεί και σκεφτόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Διότι από νομικής πλευράς κάθε μια ξεχωριστή παραβίαση προφανώς είναι η σημασίας. Κάθε υπόθεση έχει ισότιμη μεταχείριση. Όμως από οικονομικής άποψης κάποιες περιπτώσεις έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από άλλες. Εάν δούμε λοιπόν τα πράγματα σφαιρικά, θα πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε ότι οι παραβιάσεις στην αγορά της ενέργειας ή στα συστήματα των δικτύων, αυτά είναι δουλειές όπως τα λέγαμε χοντρές, είναι μεγάλες υποθέσεις, με ζουμί. Η παραβίαση λόγου χάρη σε δημόσιο διαγωνισμό για τους κανόνες της σε, στα χαρτί τουαλέτας ε, ήταν ε, πραγματικά ένα μεγάλο θέμα. Εδώ χρειάζεται λοιπόν η ανάλυση μας να είναι αυστηρή και προσεκτική. Κάτι που δεν έχει γίνει ως τώρα. Σας ευχαριστώ. Um, Mrs. I think. Κυρία Ρόιτοβα, έχουμε ακόμα χρόνο για ερωτήσεις. Έτσι καλώ ο εισηγητή μα για το επόμενο θέμα δεν έχει φτάσει ακόμα. Και την παρουσίαση του οπωσδήποτε θέλουμε να την ακούσουμε. Οπότε δεν θα περάσουμε στο επόμενο. Κυρία Ρότο, Ρόιτοβα. Και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να επανέλθουν. Κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξή. Αυτό το έγγραφο είναι άριστο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν έχει κάποια ειδική μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποια δεδομένα που λείπουν. Λόγω χάρη, αν δούμε τον πίνακα του ελέγχου ευρωστία, του fitness check, έχετε ξεχωριστά στοιχεία για την πρόοδο τη κάθε χώρα για τις τάσει που αναπτύσσονται εκεί. Διότι εδώ φαίνεται να έχουμε πληροφορίε του 2011 μόνον. Επίση θέλω να σχολιάσω ότι Ακούσαμε κάποιον από την Επιτροπή να λέει ότι αρκετές χώρες αγνόησαν την οδηγία περί υπηρεσιών. Ή τέλο πάντων δεν ενδιαφέρονται αρκετά για αυτή την οδηγία. Μα δεν το καταλαβαίνω, διότι όλες οι χώρες υποχρεούνται, υποχρεούνται να την υλοποιήσουν την οδηγία. Θα θέλαμε λοιπόν λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Κύριε Σφάμπ, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, θα ήθελα να επανέλθω κύριε Πρόεδρε σε αυτά που είπε η κυρία Ντέιλ. Σαν Επιτροπή εσωτερική αγορά, εμείς έχουμε πολλές φορές δυσκολία να αντιμετωπίσουμε αυτά που λέει η Κομισιόν, που λέει ότι είναι βέβαια σημαντική η εσωτερική αγορά και πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Όταν όμω εμεί μπαίνουμε στι λεπτομέρειε, α, λέει, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουν τα κράτη-μέλη και δεν πρέπει εμεί να επέμβουμε σε πολύ λεπτομεριακό επίπεδο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία μας απογοητεύει σε κάποιο βαθμό. Δεν είναι ικανοποιητική λοιπόν αυτή η αντιμετώπιση. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρει ποια κράτη-μέλη προχωρούν με την εφαρμογή των ρητρών της ενιαίας αγοράς και ποια όχι. Θα πρέπει η Κομισιόλα λοιπόν να μας δίνει πιο λεπτομεριακές πληροφορίες. Δεύτερον, ε, για τα θέματα των διαδικασίων επί παράβασης ε, εναντίον της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελλάδος. Νομίζω ότι το κύριο σημείο κριτικής για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς είναι ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια και δεν μπορεί κανείς να καταλαβαίνει ποιοι είναι οι, παρα... <clears throat> φορείς με τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει επαφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει παράβαση των συνδικών και επομένως θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα με αυτή την οπτική γωνία. Κυρία Ντέιλ, θέλετε να υπάρχετε το σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν απαντήσατε απόλυτα για δείκτες οι οποίοι θα βελτιώσουν την καλύτερη αντίληψή μας του επιχειρηματικού κλίματος. Μιλούσαμε με την Κομισιόν και την προηγούμενη εβδομάδα και η Αμόδιος Επίτροπος είχε τονίσει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση από την πλευρά των κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Ένα άλλο σημείο το οποίο βλέπω εδώ, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βάσει του πακέτου για τα ε, αγαθά, για τα εμπορεύματα, είχε ζητηθεί να υπάρξει ένα μονοαπευθυντικό γραφείο για τις εταιρείε που έχουν προβλήματα στην εξαγωγή αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι προεξάρχον θέμα σε αυτά που είπατε, αλλά αυτός πιστεύω ότι είναι ένας τομέας που χρειάζεται περισσότερη προσοχή για να δοθεί έμφαση στα θέματα αυτά της ε, αγοράς αγαθών. Ξέρω ότι εσείς δίνεται περισσότερη έμφαση στις υπηρεσίες, αλλά πρέπει με τρόπο ομαλό να υπάρχει μετάβαση από τον ένα τομέα στον άλλο, πιστεύω. Κυρία Ντέιλι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα του χρόνου θα έχουμε και τον δείκτη για τα αγαθά, τα εμπορεύματα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία η Γενική Διεύθυνση του Επιχειρήν θέλει να προωθήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύνδεση αγαθών και επιχειρήσεων και σύνδεση με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επόμενη ημερίδα μας θα συνδυαστεί με αυτήν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο κύριος Ταγιάννη συνεργάζεται με τον κύριο Μπαρνιέ ώστε να υπάρξει στον ατόμο μεγαλύτερη συνέργεια για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα θέματα όπως του επιχειρήν μεταξύ των νέων κοιτάζουμε τα θέματα της λεγόμενης γενιάς του 92 που τώρα είναι οι κοσάριδες και προσπαθούν να διατυπώσουν πολιτικές για τη γενιά αυτή. Σε σχέση τώρα με το πρώτο σας ερώτημα κύριε Σουάμπ, εγώ για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ασκείται τεράστια πίεση στα κρατημέλη. και οι δείκτες δεν βελτιώνονται πάντα. Στη δική μου χώρα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί και υπάρχουν μεγάλα κενά σε πολλά σημεία. Επομένως η δημόσια διοίκηση έχει πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα προτού γίνουν καλύτερα το πού ασκείται πίεση, πώ την ασκείται την πίεση και το αν αυτό θα αποδώσει καρπούς, αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι όταν κάνουμε προτάσεις προς τα κράτη-μέλη σε σχέση με το IMI ή το Solvit ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα, προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να κάνουμε τη ζωή των κρατών μελών ευκολότερη ώστε να γίνονται πιο αποδοτικά σε σχέση με το κόστος αυτά τα μέτρα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Επομένως, σε σχέση με αυτά τα στοιχεία που σας παρουσίασα, αυτά είναι αδρά στοιχεία που σας δίνουμε, αλλά αυτός είναι και ο στόχος μας. Πολλές από τις ερωτήσεις σας είναι πιο λεπτομεριακές στον α ή στο β τομέα. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες στην έκθεση για το IMI, για την παροχή υπηρεσιών κτλ. για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Αλλά μια ολιστική προσέγγιση είναι πολύ πιο σημαντική και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Επομένως, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι συμφωνώ ότι κάποιες περιοχές είναι πιο σημαντικές από άλλες, πιστεύω ότι σε κάθε κράτο μέλος υπάρχει καλή θέληση. Κάθε κράτο μέλος έχει διαφορετικό τρόπο του επιχειρήν και του εργάζεστε. Εκεί που είναι πιο εύκολο να υπάρξει συγκεντρωτική μορφή συντονισμού, να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα, όσο πιο ελαφριά είναι η διοικητική δομή, τόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει κακή θέληση. Επίση, δεν υπάρχει τίποτα πιο επιτυχημένο από την επιτυχία τη ήδη. Την ίδια. Ό,τι κάνουμε και επιτυγχάνει και γίνεται καλό για τους πολίτες και για τη δημόσια διοίκηση είναι η ιστορία επιτυχίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας το θέμα της απόσπασης εργαζομένων. <clears throat> Είναι κάτι που εισήχθη μόνο πρόσφατα στο IMI. Όλοι βλέπουν όμως ότι έχει νόημα αυτό το σύστημα και υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επομένως, αυτό είναι που προωθεί αυτές τις ε, ε, ιστοσελίδες και τις ε, δικτυακές πύλες και το IM Europe επίσης. Με, όταν με τον τρόπο αυτό κάνουμε σαφέστερο προς τους πολίτες τι δικαιώματα έχουν και τι δυνατότητες υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις γλώσσες, σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων και των πολιτών. Δύο εκατομμύρια επισκέψεις είχαμε σε ένα χρόνο. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο, αυτή είναι η πρόκληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να βγάζει νόημα αυτό που κάνουμε. Και σε σχέση με τα μόνο απευθυντικά επαφικά σημεία της επιχειρήσης και την οδηγία για τις ε, παροχή υπηρεσιών, αυτό είναι νευραλγικό και ζωτικό. Σας κατευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μας τα ξαναπείτε και για την νέα διακυβέρνηση. Θα ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μπουσουτήλ που προσήλθε για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Έχουμε την ευκαιρία με την έκθεση του κυρίου Μπουσουτήλ να συνεχίσουμε πολλά από τα θέματα που θίξαμε από τις 9. Δυστυχώς δεν ήταν εδώ από την αρχή, αλλά πάντως θα τα μάθει νομίζω αυτά που είπαμε. Λοιπόν, τώρα το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μπουζουτήλ. Είχαμε πει ότι λόγω των αλλαγών η έκθεσή του έπρεπε να καλύψει και την ετήσια έκθεση για την governance. Γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο. Έχουμε εδώ και τους σκιώδεις όχι όλους βέβαια, και εγώ είμαι από τους κοιόδης. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει εξ ονόματος της Κομισιόν η ίδια η κυρία Ντέιλι ή κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, κάποιος από εκεί θα απαντήσει. Λοιπόν, κύριε Μπουζουτήλ μου, έχετε το λόγο για το σχέδιο έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι πολύ ήθελα να είμαι εδώ πριν τι 9.45, αλλά ψήφισα σε άλλη επιτροπή. Το πολύ πούμε που έχασα την παρουσίαση. Ήταν παρανόηση. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να τα καλύψω μετά. Έχω και άλλε ευκαιρίε να συζητήσω με την Επιτροπή και θα συνεργαστώ πλήρω ε, μαζί του στο πλαίσιο τη εκθεσή μου. Τώρα η βασική ιδέα εδώ ήταν να προωθήσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς επικεντρωνόμενη στον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αλλά και με παραπομπές στην έκθεση Solvit. Η δική μου η έκθεση αρχικά σχεδιάστηκε για να απαντήσει στην 22η προσθήκη του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς που πέραν των ε, κεφαλαίων για την μεταφορά και την υλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την ενιαία αγορά στα κρατη Μας ενδιαφέρει να δούμε τις περιπτώσεις ε, επιτυχημένων αποτελεσμάτων και τις ελλειπούς, τις πλημελούς ε, μεταφοράς. Αυτά τα αποτελέσματα ήδη συγκεντρώθηκαν από πέρσι το Σεπτέμβριο, αλλά που σωστά επισημάνατε, Πρόεδρε, μετά την αρχική σύνταξη τη έκθεση, 23 τότε προσθήκη στον πίνακα αποτελεσμάτων τη εξωτερική αγορά ε, ήρθε να προσθεθεί στα προηγούμενα, όπω και το check-up τη ε, διακυβέρνηση, τη governance, μια ε, επίσης καινούργια έκθεση Solvit, οπότε με αυτές τις εξελίξεις ε, μετατρέψαμε τις προθεσμίες και το χρονικό πλαίσιο της έκθεσης αυτής, ώστε να ενσωματώσουμε και τα νέα στοιχεία. Επίσης, για να προλάβει εγκαίρως να συμβάλλει στα τελευταία αυτά ευρήματα και η δική μας η Επιτροπή. Υπ' αυτή λοιπόν τη σκοπιά κοιτάζουμε το τι αλλαγέ μπορούμε να φέρουμε στο χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή για να έχουμε έγκαιρη έγκριση τη δική μου τη έκθεση, να είναι πιο χρήσιμη και εύστοχη. Το νέο λοιπόν χρονοδιάγραμμα έχει ω εξή. Σήμερα, ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεση, προθεσμία υποβολή τροπολογιών την επόμενη εβδομάδα, 26 Μαρτίου, Δευτέρα νομίζω, το μεσημέρι, έπειτα ε, εξέταση των τροπολογιών στις 12 Απριλίου, έγκριση στην Επιτροπή 25 Απριλίου και στην Ολομέλεια τον Μάιο φέτος, στη Σύνοδο του Μαΐου. Ως προς το περιεχόμενο τώρα, το περιεχόμενο της έκθεσης. Προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο περισσότερες από τις αντιδράσεις των συναδέλφων μπορούσα, ήδη από την αρχική της εκδοχή. Συνάντησα τους ασκιώδεις εισηγητές σε μια πρώτη επαφή, αλλά και υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των οποίων η συνεισφορά και των ναι και των ΔΕ ήταν πολύτιμη. Ωστόσο, καθώς η αρχική εκδοχή της έκθεσης συντάχθηκε πολύ νωρίτερα από τον ελεγχό υγείας της τον ελεγχό της ε, διακυβέρνησης τώρα, υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα τα οποία πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις νέες εξελίξεις. Το ίδιο και για την, έκθεση, την πρόσφατη έκθεση Solvit. Η αρχική λοιπόν εκδοχή της έκθεσης επικεντρωνόταν σε δύο βασικά ε, στοιχεία. Πρώτα απ' όλα το να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά. Εδώ ε, έδωσα έμφαση στην ανάγκη τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν και να εντείνουν τις προσπαθίες τους για τη μεταφορά, αλλά και τους στόχους υλοποίησης, ιδίως εφόσον χρειάζεται καλύτερη και εγκαιρότερη ε, υλοποίηση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, καθώ αυτό είναι αποτελεσματική μέθοδο για να αντιμετωπιστεί και η οικονομική κρίση. Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης ε, έμφαση δόθηκε στα πραγματικά αποτελέσματα από την εσωτερική αγορά προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Εδώ ο αρχικός στόχος ήταν οι πολίτες να διαθέτουν λύσεις στα προβλήματα που τους δημιουργεί η εσωτερική αγορά με την σωστή χρήση των ε, ανάλογων εργαλείων και προκειμένου να καλυφθούν και οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Εδώ έπρεπε να υπάρξει μια επαναθεώρηση ώστε να δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά ακριβώ των πολιτών και όχι μόνον από τη σκοπιά του νομοθέτη, των πολιτικών εθνώντων. Έτσι λοιπόν θελήσαμε να προωθήσουμε προς τους πολίτες Μάλλον θελήσαμε να δούμε με άλλη λογική κάποιες δικές μας φιλοδοξίες που μπορεί να μην ήταν τόσο ελκυστικές για τους ε, πολίτες και τις επιχειρήσεις ή να είχαν διαφορετικές ανάγκες. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία που κοιτάξαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Και αυτά ε, τα λάβαμε υπόψη και σε σχέση με την ε, έκθεση της Επιτροπής για τον ετήσιο έλεγχο υγείας της διακυβέρνησης. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε ενδιαφέρουσα προσέγγιση, αρκετά καινοτόμο και υπέβαλε μια έκθεση που πραγματικά επικεντρώνεται στην προστιθέμενη αξία. Μάλιστα αυτό γίνεται γιατί όλα συναρμόζονται και υπάρχει μια ε, φωτογραφία, ένα πραγματικό στιγμιότυπο της πραγματικότητας που ισχύει για την εσωτερική αγορά. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλαν σκληρές προσπάθειες. Η δική μου έκθεση θα είναι μόνο το πρώτο βήμα, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τα θέματα αυτά και να επιδιώξει καλύτερο συντονισμό. Το αν θα υπάρξουν επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών της Επιτροπής και το πώς καλύτερα θα καταλάβουμε το πώς θα εφηγραμμιστούν τα διάφορα θέματα και θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στην αγορά, όλα αυτά είναι ωφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από προηγούμενες εκθέσεις που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή μας. Νομίζω αυτή τη στιγμή η σημαντικότερη προθεσμία είναι η Δευτέρα, συνάδελφοι. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών δηλαδή. Εν τω μεταξύ, καλοδεχούμενε θα είναι όλε οι προτάσει για το πώ να βελτιωθεί η έκθεση, συμπεριλαμβάνοντα τι νέε αυτέ εξελίξει που σα ανέφερα και έχοντας υπόψη ότι αυτή είναι μια έκθεση όπου γενικότερα υπάρχει συνένεση. Όλοι μπορούμε να, ε, δώσουμε, να βάλουμε το λιθαράκι μας και να ετοιμάσουμε μια έκθεση που θα είναι αποδεκτή, αποδεκτή από όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουζούτιλ. Γιατί αναλάβατε το καθήκον αυτό. Καλό θα ήταν να έχουμε μία έγκαιρη ανταπόκριση Ξέρω ότι αν και είναι καινούρια η πρόταση για τη νέα διακυβέρνηση, ήδη την αναλάβατε. Λοιπόν, τώρα τα σχόλια των γενικών εισηγητών. Ο καθηγητής Κάμπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μποσουτήλ για την έκθεσή του Νομίζω ότι κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται εδώ συνεργασία μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου και κρατών μελών που έχουν τη φυσική τάση να δρανούν και να ελαχιστοποιούν τη σημασία <clears throat> της εσωτερικής αγοράς συνήθως. Πρέπει λοιπόν να τους επιμορφώσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε βέβαια εδώ στο Κοινοβούλιο, να πληροφορήσουμε τους υπουργούς, αν και θα έπρεπε. Και ίσως θα πρέπει να συνεννοούμαστε περισσότερο μεταξύ μας οι ευρωβουλευτές. Το έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν με περιορισμένη επιτυχία βέβαια. Εγώ έχω γράψει πολλές φορές σε υπουργούς της χώρας μου η κατάσταση όπως δείχνουν οι αριθμοί βελτιώθηκε κάπως αλλά ίσως επειδή εγώ είμαι στην αντιπολίτευση μπορεί τέτοιες επιστολές μου στο μέλλον να είναι πιο αποτελεσματικές ακόμα τέλος πάντων αυτό ήταν αστείο Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για επίσημο αίτημα του Κενοβουλίου. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ αποφάσισε να το δεχτεί από τον περασμένο Φεβρουάριο αυτό το ενεκτήσιο πίνακα αποτελεσμάτων. Καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί εκτός από τη φυσική αδράνεια των χωρών μελών διστάζουν επίσης να εφαρμόσουν, να δώσουν συνέχεια σε αυτό το αίτημα. Ίσως Μία εξήγηση να είναι ότι μετά την τρομερή αύξηση των δημοσίων υπηρεσιών μετά το 60 τώρα μειώνονται και γι' αυτό δεν είναι και πιο διατεθειμένοι να εφαρμόσουν αυτά στις προτάσεις. Αλλά ο κύριος λόγος είναι η κακή και μηδενική μεταφορά της νομοθεσίας. Το δίκτυο Solvit πρέπει να ε, έχει από πιο σαφή εντολή. Γι' αυτό επιτέλους βρίσκουμε το έγγραφο για την μελλοντική λειτουργία του Solvit κάτι που το δεχόμαστε με χαρά. ίσως να χρειαστεί, ίσως να πρέπει <clears throat> να δούμε και ποια είναι τα ακόμη τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, ο συνάδελφος Μπουσουτήλ νομίζω ότι βλέπει τα πράγματα πολύ σωστά και ελπίζω να συνεισφέρω και εγώ με τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λόκεγκαρντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για ό,τι έχει κάνει τώρα δεν αποτελεί μυστικό πρόεδρε ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων, ιδίως ό,τι αφορά το Solvit, αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την ε, ομάδα μου. Για μένα, με το πέρασμα των ετών, ο πίνακας αυτός αποτελεσμάτων αποτελεσμάτων φάνηκε το πολυτιμότερο εργαλείο για να επιταχύνουμε την ε, υλοποίηση των οδηγιών όπως θέλαμε. Ε, ο επονιδισμός, ε, το naming and shaming όπως λέγεται, ήταν ένα από τα μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται. Εδώ πρέπει λοιπόν, Πρόεδρε, να φροντίσουμε όσα επισημενόνται από τον πίνακα αποτελεσμάτων να αξιοποιηθούν ώστε να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σωστά ο εισηγητή εδώ επικεντρώνεται στην έκθεση διακυβέρνηση, στην... τον ετήσιο έλεγχο υγεία. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή γιατί μας επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα σφαιρική των όσων γίνονται. Εδώ υπήρξαν πολύτιμες πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο ως προς την ίδια την έκθεση Εδώ να πω ότι δυστυχώς, και αυτό είναι μια έκφραση μιας μικρής δυσαρέσκειας, δεν έχουν γίνει πολλά ως, ε, από τα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το ποσοστό του 0,5% δεν αποτελεί πραγματική μείωση, το αντίθετο. Άρα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Ιδίω επειδή διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Γνωρίζουν πολύ καλά τα κρατημέλη τι συμβαίνει και οι δημόσιες αρχές. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Όμως, πολύ σημαντικό είναι να δοθεί και έμφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κυρίου Μπαρνιέ ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ε, ενιαία αγορά χωρίς ε, άλλες, χωρίς άλλες δυσκολίες. Η έκθεση του κυρίου Μπουζούτιλ είναι εξαιρετική, είχα την ευκαιρία να το πω και ο ίδιος και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό μέσω από τον πίνακα αποτελεσμάτων τι είναι αυτό που είναι αποτελεσματικό για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις περισσότερο, από τη δική τους την άποψη. Τα ποσοστά, ας πούμε, Κάτι που το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν επανειλημμένως. Πρέπει να τα κοιτάξουμε τα ποσοστά αυτά και να σκεφτούμε γιατί δεν μειώνονται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά, καθώς και στον δείκτη της απασχόλησης. Έχω καταθέσει σχετικά τροπολογίες και ελπίζω ότι η τελική μορφή της έκθεσης θα είναι ισόρροπη και θα εκφράζει τις απόψεις της ομάδας μου. Good. Thank you very much. Πολύ ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδης συγητές. Θα κάνω και εγώ μερικά σχόλια. Κύριε Μπουσουτήλ, ως εισηγητής και εμείς ως σκιώδης έχουμε την ε, ανάγκη να προσθέσουμε και νέο υλικό σε αυτή την έκθεση που δεν υπήρχε ακόμα όταν παρουσιάστηκε πρώτη φορά την έκθεση, αλλά είχατε προβλέψει πολλά από τα σημεία που θα ηγερθούν από τους συναδέλφους. Θα ήταν χρήσιμο για μας, πιστεύω, να εστιάσουμε περισσότερο στις ενδεχόμενες συνέργειες που έχει εντοπίσει η νέα έκθεση της Κομισιόν. Ήταν κάτι που είχαμε τονίσει πάρα πολύ στις πρώτες μας εκθέσεις, στις προηγούμενες εκθέσεις μας και στο αρχικό σας κείμενο και εσείς κύριε Μπούσουτιλ, ορθά είχατε εστιάσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα σημεία, τα μοναδικά σημεία επαφής και σύμβασης για τους πολίτες που θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο που παίζουν και τα κέντρα καταναλωτών σήμερα στην Ευρώπη. Το είχα αναφέρει λοιπόν αυτό, προτού αναφερθήκατε, προτού αναφερθείτε στην ενιαία αγορά για τα εμπορεύματα που πρέπει και αυτή να συμπεριληφθεί. Και αυτό ήταν τμήμα του τις δέσμες μέτρων για τα αγαθά. Αλλά έχει κάπως εξαφανιστεί προς το παρόν και πρέπει να το επαναφέρουμε σε κοινή θέα. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει αναφέρει πολλά χρήσιμα πράγματα στην έκθεση ευκυβερνησίας για τις συνέργειες. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά φιλόδοξη η αντιμετώπιση της Κομισιόν και ίσως και εκεί θα πρέπει να τους πιέσουμε λιγάκι. Ένα περαιτέρω σημείο το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό, αλλά το οποίο είναι και ενωφανές και σε αυτή την έκθεση, είναι το διάγραμμα κλειστού βρόχου που παρουσίασε η κυρία Ντέιλι στην αρχή. Πώς τα δεδομένα λοιπόν τα οποία συλλέγονται από όλα αυτά τα σημεία επαφής αποτελούν και ένα σημαντικό πόρο για μας και για άλλους λήπτες αποφάσεων για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε <clears throat> αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Και βλέπω ότι στην ε, επισκόπηση της έκθεσης αυτής αναφέρεται το θέμα της ε, σύνδεσης με την έκθεση για τα επαγγελματικά προσόντα και το θέμα της αμοιβαία ε, ε, αξιολόγησης στην οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Έχουμε λοιπόν εκεί πέρα πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά σχόλια, σημαντική ανάδραση που μπορούμε να αποσπάσουμε από αυτή την επισκόπηση και μπορούμε να τα κοιτάξουμε αυτά και πρέπει να τα κοιτάξουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια. Χρειαζόμαστε επίσης ανάδραση από την εφαρμογή του πακέτου για τα αγαθά και για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο λοιπόν και από εκεί να αποκομίσουμε πληροφορίες. Για μένα λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ θετικό, Σίμων, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα νέα στοιχεία της έκθεσης ευκυβερνησίας που έχουν να κάνουν με συνέργειες και να τα ενσωματώσει στην έκθεσή σου, γιατί αυτό θα ενισχύσει και θα κάνει ιδιαίτερα ισχυρή αυτή την έκθεση. Και τέλος έχω να κάνω και κάποιες προτάσεις τροπολογιών σε σχέση με αυτά που ανέφερα στην κυρία Ντέιλι προηγουμένως. Θα πρέπει να βρούμε κάποιους δείκτες απόδοσης σε σχέση με την ε, συνειδητοποίηση των επιχειρήσεων και των πολιτών, ιδίως των τελευταίων, για το πώς μπορούν να αποκομίσουν πληροφορίες και επίσης συνειδητοποίηση από την πλευρά των επιχειρήσεων αν έχουν πραγματικά αντίληψη των ευκαιριών που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά και αν γνωρίζουν τα μονοπευθυντικά σημεία επαφής. Μπορεί να έχει αυξηθεί ο αριθμός των σημείων επαφής σε σχέση με τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να υποφεληθούν από την ενιαία αγορά ή σε σχέση με αυτούς που ενδιαφέρονται για προγράμματα καταναλωτών ή οτιδήποτε τέτοιο, εξακολουθούν να είναι πολύ λίγα αυτά τα σημεία τα σημεία επαφή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα πιο πολλά σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά είναι μόνο 1.400, όχι 1.800 όπως είπα προηγουμένως, στο Ηνωμένο Βασίλειο. <clears throat> Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια μέτρα απόδοσης στα κράτη-μέλη, κάποιο τρόπο να καταμετρήσουμε την απόδοση στα κράτη-μέλη και πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι πάρα πολύ εστιασμένα και σοβαρά στο να εφαρμοστούν όλα αυτά. Άλλα μέλη, κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσουτήλ για το πολύ καλό σχέδιο έκθεσή του. Θέλω να σταθώ τώρα σε τρία σημεία, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία αναφέρθηκαν και από τον κύριο Μπουσουτήλ. Το πρώτο είναι ο βαθμός μεταγραφής των οδηγιών και εφαρμογής τους στα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από το δικό σα κείμενο. Είσαστε μάλλον διπλωματικό και αυρόφρον σε αυτά τα οποία λέτε. Αλλά παραδείγματο χάρη μπορούμε να αναφέρουμε την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Όταν ήμασταν στο τριγωνικό διάλογο με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, είχαμε τότε ζητήσει από το Συμβούλιο των Υπουργών να έχουμε κάπω μακρότερε προθεσμίε ακριβώ για να μπορούμε να έχουμε την αμοιβαία αξιολόγηση και άλλους τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Και είπανε πολλά χρόνια, τα οποία είπαν ότι θέλουν δύο χρόνια και όχι δυόμιση ή τρία χρόνια. Αλλά τα κάτι μελη τα οποία είχαν μια τέτοια άποψη, όταν το θέλουν αυτό, θα έπρεπε να περιμένουμε από τα κάτι μελη ότι θα είχαν κάνει αυτήν την εφαρμογή της οδηγίας. Και όχι να πρέπει να τα οχλούμε και να πούμε ότι πρέπει αυτά να σεβαστούν τις ίδιες τις αποφάσεις τους και να τηρήσουν τα υπεσχημένα από αυτούς. Ένας δεύτερος τομέας που θέλω να υπενθυμίσω είναι το Solvit. Έχουμε συζητήσει διαμακρών για το Solvit και αυτό είναι θετικό. Γιατί είναι μεγάλος ο τομέας που καλύπτεται από το Solvit, αλλά θα έπρεπε, πιστεύω, και αυτό το αναφέρατε, κύριε Μπουσουτήλ, να σκεφτούμε περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να δημιουργηθούν τα σημεία επαφής για το Solvit. Πριν από 1,5 χρόνο ήμουνα στο Παρίσι και είδα εκεί τα γραφεία του Solvit και διαπίστωσα, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο κάποιοι ασκούμενοι εργαζόντουσαν στα σημεία αυτά του Solvit. Δεν πρόκειται λοιπόν μονάχα για τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτά τα γραφεία, αλλά δεν λέω ότι είναι θέμα ποιότητα. Ακόμα και οι ασκούμενοι μπορεί να έχουν υψηλή ποιότητα, αλλά το επίπεδο εμπειρία που έχουν και η ικανότητά του να παίρνουν πολιτικέ αποφάσει, <clears throat> οι οποίε είναι σημαντικού χαρακτήρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να προσθεθεί στην έκθεση, λοιπόν, πιστεύω, κύριε Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Θυμάμαι το σημείο αυτό που αναφέρατε κυρία Γκέπχαρτ, την παρατήρησή σας για το γραφείο των Παρισίων της Λουτιτίας, γιατί θυμάμαι ότι το είχατε πει στον Γάλλο εκπρόσωπο όταν ήμασταν εδώ σε μια κρόαση. Κανονικά υπάρχει ένας ε, εκπρόσωπος από τη Γαλλία που παρακολουθεί τις συνεδριάσεις μας και θα το σημειώσει πιστεύω. Κυρία Ρούλα, τώρα εσείς θέλετε να πείτε κάτι ως ε, σκιώδης εισηγήτρια. Όχι, δεν θέλετε. Κάποιος άλλος πρωτού δώσει το λόγο πάλι στην Κομισιόν. Όχι. Ποιο θα λάβει το λόγο λοιπόν από την Κομισιόν, γιατί έχουμε πολλού από την πλευρά τη Κομισιόν. Κύριε Ντέιλι. Κάνουμε μια μάχη μεταξύ μα. Αποφασίστε, ξεκινήστε εσεί ω επικεφαλή τη ομάδα. Έχουμε τέτοιο ενθουσιασμό που δεν κρατιόμαστε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουσοτήλ Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ασχολείστε με αυτό το θέμα, διότι η δική μας η ανάλυση έχει ω εξή. Ο άνεμος είναι όριο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τον Ιούνιο να υπάρξει έκθεση από την Επιτροπή για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ευκυβερνησία στην εσωτερική αγορά. Ήδη από τον Ιούνιο λοιπόν έχουμε αυτή την προτροπή, το δικό σας το έργο σήμερα και οι ιδέες που συνεισφέρετε με την έκθεσή σας, καθώς και το επίπεδο φιλοδοξιών που εκφράζει, είναι σημαντικά, διότι θα μας βοηθήσουν να έχουμε επιχειρήματα και να προχωρήσουμε. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς την ΙΜΚΟ. Πρέπει να το πω αυτό. Εσείς είστε κάτι σαν άγγελος φύλακας για μας σε αυτά τα θέματα. Όσο περισσότερα κάνετε εσείς, τόσο περισσότερο μας πρόχνετε και εμάς προς τα μπρος. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, εάν ετοιμάσετε κάτι που θα δημοσιευτεί, θα το έχουμε στα χέρια μας το Μάιο, αυτό είναι πραγματικά τέλειο. Θα προλάβουμε να το λάβουμε υπόψη σε σχέση με όσα θα συμπεριλάβουμε στην ε, ανακοίνωσή μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, εκ παθέων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να είμαστε φυλακά άγγελος για την εσωτερική αγορά γενικότερα. Ελπίζουμε να γίνει και αυτό. Υπάρχει μια όσμωση εδώ τη δουλειά μα με την Επιτροπή. Παρόλο που εσεί διατηρείτε το δικαίωμα πρωτοβουλία, υπάρχει αυτή η διαρκή επικοινωνία μεταξύ μα. Υπάρχουν άλλα σημεία που θέλετε να σχολιάσετε εσείς οι συναδελφοί σας. Ναι, να απαντήσω για τον πίνακα αποτελεσμάτων πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε να μελετήσουμε την έκθεση αυτή, όχι μόνο όμω αυτή. Διότι έχει ετοιμάσει πάρα πολλέ εκθέσει ήδη η ΕΜΚΟ για τους πίνακες αποτελεσμάτων. Και ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα προχώρησαν παράλληλα. Πολλές προτάσεις τη ΕΜΚΟ ήδη έχουν συμπεριληφθεί και ληφθεί υπόψη. Στου πίνακε αποτελεσμάτων. Ίσως να προχωρήσουμε και παραπέρα. Όμω, ο πίνακο αποτελεσμάτων σε αυτή την περίπτωση αποτελεί ένα, μια βάση. Οι εκθέσει σα μα δίνουν ευκαιρίε να σκεφτούμε παραπέρα, περαιτέρω. Να προσθέσουμε νέε πτυχέ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Μπουσούτελ για την προθυμία του, για τι συζητήσει που είχαμε τώρα και για τεχνικά θέματα. Γιατί ο πίνακα αποτελεσμάτων έχει ιδιαίτερα τεχνικέ πτυχέ κάποιε φορέ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια από τις τέλειες ευκαιρίες να προχωρήσουμε τη σκέψη μας στα θέματα αυτά. Κάποιος άλλος για το Solvit, για κάτι ανάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς μια πληροφορία για το γαλλικό γραφείο Solvit. Έχει βελτιωθεί πολύ έκτοτε. Έχουν δύο μόνιμους υπαλλήλους πλέον σε εκείνο το γραφείο, που είναι αρμόδιοι και για άλλα ζητήματα βεβαίως, όχι μόνο για το Solvit αλλά έχουν ακόμη μεγάλο φόρτο εργασίας. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, περαιτέρω στελεχώσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι ασκούμενοι, οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι η κυρία Γκέμπχαρτ χαίρεται ιδιαίτερα. Κύριε Μποζούτιλ, θέλετε να ε, συνοψίσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που τόσο ενεργά συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και τους ευχαριστώ και για τα ευγενικά τους λόγια. Πρόεδρε, πριν αρχίσει εδώ αυτό που κάνουμε να φαίνεται σε μια ανταλλαγή επένων μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι εάν υπάρξει ο προγραμμικό λόγο να επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα το παραλείψω. Σε αυτή την περίπτωση, περισσότερο μα ανησυχούν όμω εδώ τα κράτη-μέλη παρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα μα απασχολούν το τι μέρημνε, τι προτεραιότητε έχουν οι πολίτε, οι επιχειρήσει. Και να σταθώ σε δύο σημεία που θεωρώ ότι είναι τα πλέον σημαντικά που ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Πρώτον, το θέμα τη υλοποίηση. Είμαι 100% βέβαιο, συνάδελφοι, και απευθύνομαι ιδίω σε εσά, κυρία Γκέπχαρτ, ότι στον πίνακα αποτελεσμάτων τη εταιρική αγορά επικεντρωνόμαστε βεβαίω σε μεγάλο βαθμό στην μεταφορά, αλλά να φτάνουμε στην υλοποίηση. Ακόμη μένουμε να κοιταζόμαστε μεταξύ μας με ανοιχτά τα στόματα, χωρίς να υπάρχουν επαρκή αποτελέσματα. Κάποια κράτη-μέλη έχουν μια συγκεκριμένη στάση ως προς την υλοποίηση που είναι παράξενη. Είναι σαν να λένε, εντάξει, μεταφέραμε τους νόμους, Θέλουμε και θέλετε και να τους υλοποιήσουμε τώρα. Αυτή τη στάση θα πρέπει να την ε, πατάξουμε. Θα πρέπει να την πατάξουμε διότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τη μεταφορά, αλλά εν τέλει με το τι γίνεται με την πραγματική υλοποίηση. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ, το οποίο το, το σχολιάσατε εσείς κύριε Πρόεδρε, είναι το ενιαίο σημείο επαφή, το μοναπευθυντικό αυτό σημείο. Εγώ είμαι μέλος και της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίο που λαμβάνουμε πρόσφυγες απευθείας από τους πολίτες. Εάν δει κανεί τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς από τη σκοπιά των πολιτών, δηλαδή των αναφορών που υποβάλλουν, είναι σαν να κοιτάζουμε το ίδιο ακριβώς θέμα, αλλά από τελείω διαφορετικό σημείο. Πρέπει να πω ωστόσο, και νομίζω ότι και εσείς πρόεδρε έχετε κάποιο, κάποια συμμετοχή εδώ, ότι καλό είναι να ε, συνδυάσουμε τις προοπτικές της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς όταν μιλάμε για τη σημασία του ενιαίου σημείου επαφής. Εν τέλει, οι πολίτες δεν γνωρίζουν κάποιες φορές. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γνωρίζουν από μόνοι τους με ποιον να έρθουν σε επαφή όταν κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα τους απασχολεί. Εμείς θα πρέπει να του διευκολύνουμε. Εμείς θα πρέπει να προβάλλουμε το ενιαίο σημείο επαφή και αυτό είναι ζωτική σημασία. Νομίζω ότι το Your Europe, αυτό το πρόγραμμα, η Ευρώπη σου, είναι ένα τεράστιο βήμα πρόοδου. Ελπίζω όμως ότι θα το προωθήσουμε ακόμη περισσότερο. Συμπερασματικά, περιμένω τις τροπολογίες με ανυπομονησία και όποιος συνάδελφος θέλει να συζητήσουμε και ακόμη και στο γραφείο μου τις τροπολογίες διμερώς, ευχαρίστω για να φτάσουμε σε συνένεση. Μην ξεχνάτε ότι η προθεσμία είναι πολύ κοντά, τη Δευτέρα κιόλα. Πάντω, τα γραφεία των σχεδόν εισηγητών έχουν ήδη δείξει ιδιαίτερη συμμετοχή στην εκθεσή μου. Οπότε δεν νομίζω τώρα να προκύψουν ζητήματα μείζωνος σημασίας που να μας εμποδίσουν να ολοκληρώσουμε. Να καταλήξουμε τέλο πάντων σε συνένεση. Ανυπομονώ λοιπόν για τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Well, thank you very much indeed for your work on that. Ευχαριστούμε. Απλώ να θυμίσω σε όλου ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών τη Δευτέρα το μεσημέρι θα ακολουθήσουμε το νέο χρονοδιάγραμμα όπω είπαμε. Και από όσα είπε η κυρία Ντέιλ είναι φανερό γιατί χρειάζεται από το νέο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ την κυρία Ντέιλ και την ομάδα τη που ήταν μαζί μα σήμερα το πρωί. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες ακριβώς στις 10.30, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας, εάν όχι να τις πάρετε από τα γραφεία σας, στον αμέσως από κάτω όροφο. Και στις 10.30 θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Μπίλαν, νομίζω είναι η πρώτη. Uh, uh, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία για αυτούς που έχουν μόλις έρθει και για αυτούς που μας βλέπουν από το διαδίκτυο. Έχουμε αλλάξει λιγάκι το χρόνο διάγραμμα για σήμερα το πρωί. Αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Κόμης. Σήμερα θα ψηφίσουμε πρώτα. Μήπως μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία και λιγότερη βαβούρα, παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση Μπίελον για την διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς και μετά θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του κυρίου Έγγελς για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας για να κάνει κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και οι σκιώδει μπορεί να θέλουν να κάνουν σχόλια πριν από την ψηφοφορία, αλλά πρώτα εσεί κύριε Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε στη χθεσινή μας συνεδρίαση τη συμβαστική τροπολογία, είχαμε μια μακρά συζήτηση για τα θέματα αυτά. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και, και τα μέλη της γραμματείας για τη βοήθειά τους στην έκθεση αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που με τη βοήθεια του Θεού θα ψηφίσουμε σήμερα. Κάποιο άλλος θέλει να λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των σκιωδών εισηγητών του ΕΛΚ, των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα της προστασίας δεδομένων. Πρέπει να κρατάμε λοιπόν τα δεδομένα μονάχα όσο χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του συστήματος EMI ή IMI. Και επειδή ζητάμε από την Κομισιόν να διευρύνει αυτό το σύστημα για σημαντικά θέματα και επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να αξιολογήσουμε τις ε, επιπτώσεις της τροποποίησης της αρχικής πρότασης της Κομισιόν όπως ζητάει ο εμείς θα υποστηρίξουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν 18 μήνες για το μπλοκάρισμα και 5 χρόνια για την διαγραφή. Ζητήσαμε λοιπόν από τη Γραμματεία να μας δώσει και περαιτέρω στοιχεία. Θέλουμε να παραμείνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί στο να αναθεωρήσουμε την άποψή μας για το χρόνο διατήρηση των στοιχείων αν η εμπειρογνωμοσύνη μα δείξει άλλη κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεδομένου ότι οι συνολικοί κανονισμοί για την ε, προστασία των δεδομένων είναι υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητα μεταξύ τη δική μα απόφαση και τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ζήτησα σε διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία και μια γνώμη, μια γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά για να συνδυάσουμε τα δύο αυτά στοιχεία. Άλλα σχόλια πριν ψηφίσουμε. Όχι, πάμε να ψηφίσουμε τότε. Θα χρησιμοποιήσω τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θέλω οι εισηγητές των δύο μεγάλων παρατάξεων, η κυρία Γκέπχαρ και ο κύριος Φαμπ, να μου δείχνουν ποια είναι η κατεύθυνσή του σε κάθε τροπολογία. Τροπολογία 8 του ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έχουμε ένα σύνορο, ένα μπλοκ τροπολογιών. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 9. Το αντίστοιχο τμήμα 2 της τροπολογίας 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 50. Γκρέχ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεκτή 51 κάρας υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή πάμε στην τροπολογία 61 Λόκεγκαρ. ψήφι υπέρ κατά Α, δεκτή 63 Πάξας υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 της κυρίας Ρούλα ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται 15 του εισηγητή υπέρ κατά δεκτή 16 του εισηγητή υπέρ κατά δεκτή 17 Δεύτερο τμήμα του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 18 Μπίλαν υπέρ κατά γίνεται δεκτή. 19 υπέρ κατά δεκτή. 20 με προφορική τροποποίηση του κυρίου Μόρτεν Λόκεγκαρτ με την προφορική τροποποίηση που αναφέρει υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκπίπτει 20 κατά συνέπεια. 66 και 67 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 21 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68 τριανταφυλλίδι υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται και αυτή. 70 εκπίπτει το επόμενο μπλοκ εκπίπτει. Πάμε στην 23 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 75. Τριανταφυλλίδης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 μπίλαν υπέρ κατά απορρίπτεται 76 76 όχι 26 όπως είπα με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 και 74 εκπίπτουνε 26 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 77. de Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 27, 28 και 29 από κοινού συλλήβδιν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 78 σε τμήματα της κυρίας Ρούλα. Με χωριστή ψηφοφορία τμήμα 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Μπίλεν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79. 30 φιλίδης. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 79. Πέρας. Απορρίπτεται 15-17. Τροπολογία 80. Ρούλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Ρίλε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 82 Λόκεγκαρτ υπέρ κατά δεκτή 31 του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται 83 Ριουλε, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Πέρας. Δεκτή. 24-11. 84. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 85. Ρίλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 86. Ρίλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε στην 33 του εισηγητή για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 90 30 φιλίδης υπέρ κατά απορρίπτεται 34 του εισηγητή ελέγχω αν εκπίπτει δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε 35 Μπίλαν υπέρ κατά απορρίπτεται 36, 37, 38 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε 39 μπίλαν υπέρ κατά απορρίπτεται 91 ρούλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 ρούλα υπέρ κατά δεκτή 40 μπίλαν ε, δεν χρειάζεται πάλι να την ψηφίσουμε, συνδέεται με προηγούμενες ψηφοφορίε. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. 41. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 42. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα. 43. Κρέχ αν αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απέριπτε. Ε, δύο και τρία πάλι εξαρτώνται από προηγούμενες ψηφοφορίες. 44 Σάλτε υπέρ, κατά, δεκτή. 4 έχει αποσυρθεί, 45 Κοράτσα Μπίλτ και άλλοι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 46 εκπίπτει τροπολογία 5 υπέρ κατά απορρίπτεται 47 ρίλε υπέρ κατά δεκτή 6 του εισηγητή υπέρ άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 6 του εισηγητή Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς. 25-11. 48. Κορατσαμπίλτ υπέρ. Κατά. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 7 εξαρτάται από προηγούμενες τροπολογίες. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της ε, έκθεση όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 36-0. Συγχαρητήρια. Με μία αποχή. Μία αποχή. Του κυρίου Ντε Κύριε Μπίλαν, θέλετε να πείτε κάτι για την ε, ψηφοφορία. Ναι, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την έγκριση της έκθεσης. Θα ήθελα όμως επίσης να σας ζητήσω την εντολή να αρχίσω διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Μάλιστα, πρέπει όμως να συμβουλευτώ τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων αν θέλουν να αρχίσει τώρα η διαπραγμάτευση, να την εγκρίνουμε δηλαδή ή αν πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα οι συντονιστές. Αν είναι εδώ οι συντονιστές συμφωνούν, να δώσουμε την εντολή στον εισηγητή να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Πρόεδρε, γενικά είμαστε υπέρ. Και αφού το είχαμε αποφασίσει στους συντονιστές, συμφωνούμε και τώρα. Εντάξει, θα ψηφίσουμε και επίσημα, αλλά να ακούσω τις απόψεις των συντονιστών και συντονιστριών. Κυρία Γκέπχαρτ. σε αυτήν την περίπτωση και η δική μου ομάδα θα συνενέσει να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία γιατί ήταν σαφές το αποτέλεσμα και από ό,τι γνωρίζω και το Συμβούλιο δεν απέχει στην απόψή του από τη θέση του Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια μακρά και ε, εργόδη διαδικασία και εμείς συμφωνούμε λοιπόν να δοθεί εντολή στον εισηγητή. Κύριε Μάντες. Ούτε εμείς έχουμε πρόβλημα. Ούτε εμείς. Η κυρία Ρούλα τα ίδια. Ωραία λοιπόν. Τότε ψηφίζουμε την πρόταση να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, να δοθεί εντολή στον κύριο Μίλαν εξ ονόματος της Επιτροπής μας να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση διανατάσεως της χειρός. Α, όχι, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη χορήγηση της εντολής. Λίγοι. Λοιπόν, 35 ομοφωνία. Είναι σαφής η εντολή. Ήταν κανείς αντίθετος και δεν δούλεψε το μηχάνημα. Όχι, λοιπόν, ναι ευχαριστώ πολύ λοιπόν, ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Σαφές το αποτέλεσμα. Κύριε Βίλαν, θέλετε να προσθέσετε τίποτε άλλο. Όχι, όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ήδη κάνει μερικές πρώτες επαφές με την Δανική Προεδρία και προβλέπω και άλλες στις 11 Απριλίου. Να καταλήξουμε λοιπόν υπό την Δανέικη Προεδρία. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ για αυτόν τον ρόλο που παίξατε. Τώρα η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση Έγγελ για το κοινό σύστημα φορολόγησης των ιών. Θέλετε να σχολιάσετε τίποτα προηγουμένως κύριε Έγγελ. Όχι, τίποτα ιδιαίτερο. Ίσως απλώς να ξαναπούμε το, αυτό που είναι προφανές, δηλαδή ότι δεν θα είναι ίδιο το αποτέλεσμα με το προηγούμενο, γιατί υπάρχει διχογνωμία. Ό,τι και να ψηφίσουμε όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Παρόλα αυτά, αν εγκρίνουμε αυτά που προτείνω, νομίζω ότι θα έχουμε συμβάλει στην πρόοδο του θέματος το οποίο θα μας συνοδέψει για πολύ καιρό ακόμα. Any of the shadows was uh, Μάλιστα. Ο κ. Μάντες είχε ζητήσει το λόγο. Απλώς να δηλώσω ότι θα τα καταψηφίσουμε όλα. Γιατί δεν συμφωνούμε με χωρίς τι πρόταση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Έγκελ για τη δουλειά του, αλλά ως θέμα αρχής τα καταψηφίζουμε όλα, όχι σε όλα. Γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτή τη χωριστή πρόταση για τον φόρο των δοσαληψιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις γύρισα από την Επιτροπή Οικονομικών που η πρόεδρος είναι γυναίκα και γι' αυτό κόντεψα να σας πω κυρία πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Έγγελ για όσα έχει κάνει. Φυσικά η δική μας θέση είναι λίγο διαφορετική. Γενικά όμως συμμερίζομαι τη θέση του κυρίου Μάντερς, δηλαδή ότι αν δεν είναι σφαιρικός αυτός ο φόρος μπορεί να βλάψει τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν πιστεύουμε ότι ο τομεύς αυτός πρέπει να τιμωρηθεί για την κρίση. Ευχαριστούμε. Um, Πολύ αστείο κύριε Πρόεδρε. Ίσως οι συντηρητικοί τώρα να λυπούνται, να εκφράζουν τη λύπη τους γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τα πράγματα. Το καταλαβαίνω, αλλά αποσιοποιητικά. Ο καθηγητής Κάμπος για τους ακριβώς αντίθετους λόγους εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή. Δεν είναι τιμωρητική, είναι διορθωτική. Είναι ένας τρόπος να βελτιωθούν τα οικονομικά και να γίνει, εξισορροπηθεί πιο δίκαια η κατάσταση. Μάλιστα, ωραία, είπαν όλοι τις θέσεις τους. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Ορίστε. Λοιπόν... Τροπολογία 31 με την προφορική της αλλαγή υπέρ, κατά, yes, εγκρίνεται. 31 καταπίπτει. 32 του καθηγητού de campus υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Α, όχι, θα την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά η 33. Ηλεκτρονικά έληξε απερίφθη 18 είναι υπέρ γιατί κάποιος δεν είχε την κάρτα ναι. λοιπόν απορρίπτεται πάντως 18-19 35 του κυρίου Πάκσας υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 34 καταπίπτει, 36 υπέρ κατά απορρίπτεται. 37 de Jong υπέρ κατά απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 για ένα 3β νέο ηλεκτρονικά 40 έληξε απορρίπτεται 41 υπέρ κατά απορρίπτεται Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48 της κυρίας Γκάου Πέλτς υπέρ κατά που 49 του καθηγητού Ντε Κάμπους υπέρ κατά εγκρίνεται 50 υπέρ κατά εγκρίνεται 51 άρα καταπίπτει 52 De Jong υπέρ όχι ηλεκτρονικά για την 52 ηλεκτρονικά έληξε απορρίπτεται πανηγυρικά 9 του εισηγητού υπέρ κατά εποχές 53 υπέρ όχι ηλεκτρονικά την 53 ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά. Έληξε. Απορρίπτεται. 54 De Γιόγκ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 De Γιόγκ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. 56 καταπίπτει. Οι 57 και 58 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 11 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Χέρ εγκρίνεται. 12. έχει καταπέσει. Γιατί εγκρίθηκε η 9. 13 και 14 καταπίπτουν 15 με προφορική τροποποίηση που βλέπετε στα χαρτιά υπέρ κατά εγκρίνεται η 14 ήταν αυτή 15 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται τώρα 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 ηλεκτρονικά. Έλεξε. Απορρίπτεται 20 του εισηγητή με προφορική τροποποίηση που βλέπετε εδώ στα χαρτιά σας υπέρ κατά αν εγκρίνεται 20 έχει καταπέσει 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά απορρίπτεται 1 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 23 υπέρ κατά απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπάρχει μια αλλαγή νομίζω εδώ ότι υπάρχει θα ήθελα πρώτα την παράγραφο χωρίς την έκφραση κράτη-μέλη, η οποία θα ψηφιστεί χωριστά. Καταλάβατε όλες. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα χωρίς το member states υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα οι λέξεις κράτη-μέλη υπέρ κατά απορρίπτεται 27 de Jong υπέρ κατά απορρίπτεται. 3 του εισηγητή υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 4 του εισηγητή υπέρ, κατά 5 υπέρ κατά Δε, 30. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έληξε. Απορρίπτεται. Τώρα το σύνολο της νομοδότησης άρχεται ηλεκτρονικός. Έληξε. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, 28 μάλλον, 8 κατά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Έγγελ για όλα όσα κάνατε για μας. Ελπίζω να διασκεδάσετε στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή με τη γνωμοδότησή μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. So now we're going to move να περάσουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γκέπχαρτ. Παρακαλώ όμως, επειδή έχουμε ακόμη δουλειά, όποιοι δεν θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, ας φύγουν ήσυχα. Θέλουμε κυρία Γκέπχαρτ να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στους φακέλους σας, αλλά πρέπει να έχετε λάβει ήδη το αντίγραφο. Αυτή θα είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε μετά την επίσημη απόφαση της συνδιάσκεψης των Πρόεδρων να απορριφθεί το έτοιμά μας για κοινή έκθεση με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Πολεμήσαμε σκληρά εκ μέρους της κυρίας Κέπχαρ γι' αυτό, δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα είναι καθήλυνα αρμόδια, αλλά και η κυρία Γκέπχαρτ συνεργάζεται στενά με τον εισηγητή και νομίζω μπορούμε να περιμένουμε ότι θα επηρεάσει αρκετά η έκθεσή μας στην την τελική έκβαση. Ας μας τα εξηγήσει αυτά η κυρία Γκέπχαρτ παρουσιάζοντας την πρότασή της. Γνωρίζω ότι έχει αλλάξει το πρόγραμμα για όλους σας, οπότε θα ήθελα να δω πόσοι από τους συζητητές είναι εδώ, ο κύριο Ο κύριος Σμιτ θα έρθει, ο κύριος Μάντερς. Ο κύριος Σμιτ έρχεται ή θα μιλήσετε εκ μέρους του. Α, νάτος. Δεν σας είδα. Ο κύριος Σμιτ, η κυρία Τουρούνεν, ο κύριος Ντεγιόγκ. Εγώ θα εκφράσω την άποψη του κύριου Φόξ, δεν μπορεί να είναι εδώ. Νομίζω ο κύριος Πελέ είναι εδώ από την Επιτροπή. Χωρίς καθυστερήσεις λοιπόν. Το λόγο έχει η συγκεκριά μας, κυρία Γκέπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κρίμα που η συνέλευση των Πρόεδρων αποφάσισε να απορρίψει την ε, αίτησή μας για συν, συναπόφαση των δύο επιτροπών και είπε ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή που είναι η αρμόδια επί Είναι ένα θέμα λοιπόν που έχει να κάνει με τα θέματα των καταναλωτών και έπρεπε και εμείς να έχουμε ισότιμη μεταχείριση. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω όσο μπορώ να δώσω μεγάλη ορατότητα στην έκθεση της ε, Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα των καταναλωτών. Ουσιαστικά θα έχουμε μια μορφή ενισχυμένης συνεργασίας, επομένως η Επιτροπή μας θα εμπλακεί πλήρως στη συζήτηση αυτής της έκθεσης. Τίθεται εδώ ένα θέμα που είναι θέμα προστασίας των καταναλωτών όταν μιλάμε για το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να καλύψουμε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τους καταναλωτές με τη στενή έννοια της, του όρου, αλλά και μικρές επιχειρήσεις, φοιτητές, και άλλα άτομα τα οποία πρέπει να αποκτήσουν πλήρω αυτό το δικαίωμα πρόσβασης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν θέμα να έχουμε ένα σαφή ορισμό σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω το εξής. Έχω τονίσει ήδη και στο παρελθόν ότι θα πρέπει κανείς να μην θεωρήσει ότι υπάρχει υποχρέωση των πολιτών να έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Εγώ δεν έχω πει τίποτα τέτοιο. Ο πολίτης μπορεί να θέλει να κρατήσει τα λεφτά του κάτω από το στρώμα του. Δεν είναι θέμα καθήκοντος του πολίτη. Αλλά είναι το δικαίωμα να έχει κάνει ένα τραπεζικό λογαριασμό ακόμα και ανέαστεγος. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ακόμα και οι άστεγοι μπορεί να έχουν φόβο να τους ληστέψουν στο δρόμο, εκεί που κοιμούνται, και θα ήταν πολύ καλό για αυτούς να έχουν το δικαίωμα να έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Είναι επίσης το θέμα των φοιτητών που με το σύστημα Εράσμους με άλλο τρόπο σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα, από τη δικιά τους χώρα, θέλουν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, αλλά δεν μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν λοιπόν μια τράπεζα τους λέει ότι δεν μπορείτε να έχετε ένα λογαριασμό, επειδή δεν έχετε μια διεύθυνση. Δεν θέλω λοιπόν οι νέοι να έχουν αυτή την αντιμετώπιση της Ευρώπης ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός σε εθνικά συστήματα και δεν υπάρχει κάτι το ενιαίο. Λένε ορισμένοι ότι υπάρχει το σύστημα ΣΕΠΑ, αλλά αυτό δεν λειτουργεί πλήρως. Επομένως πρέπει μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα να υπάρξει μια λύση για να μπορεί όλος ο πληθυσμός της Ευρώπης να έχει πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Και σε αυτό το δικαίωμα πρόσβαση περιλαμβάνονται και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με ένα βασικό λογαριασμό. Κάθε άτομο που βρίσκεται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί πληρωμές μέσα από αυτόν τον ε, λογαριασμό, να μπορεί λοιπόν να ανοίγει και να διαχειρίζεται ένα τέτοιο βασικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από τον έχει κάποιο άλλο λογαριασμό σε ένα άλλο κράτο μέλο ή όχι. Γιατί σα είπα το παράδειγμα των φοιτητών, οι οποίοι ίσω σε κάποιο διάστημα θα πρέπει να παραμείνουν σε μια άλλη χώρα, μπορεί να έχουν ένα λογαριασμό στη δική του χώρα μέλη, αλλά πρέπει να έχουν και την ευκολία να ανοίξουν λογαριασμό στο κράτο μέλο όπου σπουδάσουν. Τα κάτι μέλη λοιπόν θα πρέπει να πάρουν τι απαραίτητε πρόνοιε, και γι' αυτό τονίζω ότι εδώ είναι θέμα των κρατών μελών και όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει η δυνατότητα πρόσβασης <clears throat> σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και να είναι δυνατόν για τον καταναλωτή να έχει απόλυτη ε, πληροφόρηση για το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο λογαριασμό και επίσης να έχει την απαραίτητη νομική αρρωγία να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν περιπτώσεις στι οποίε μπορεί να μην δοθεί μια τέτοια πρώτα πρόσβαση στον καταναλωτή, αλλά αυτό θα πρέπει να αιτιολογηθεί σαφώς και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ένα θέμα που είδαμε και σε άλλους τομείς, όπως είναι το ξέπλυμα χρημάτων ή σε καταστάσεις οι οποίες είναι ασαφείς, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι έχουν πάντα αυτές τις δυνατότητες να πούν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού λογαριασμού, αλλά θα πρέπει να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει άρνηση δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού μόνο σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με καταπολέμηση διαφθοράς, ξεπλήματος χρημάτων ή για θέματα εθνικής ασφαλείας. Μόνο μέσα σε τέτοια <clears throat> πλαίσια φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια άρνηση για τη δημιουργία ενός τραπεζικού λογαριασμού. Μετά από πολλές σκέψεις έχω καταλήξει επίσης στο συμπέρασμα ότι τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέψουν ότι όλες οι τράπεζες που έχουν ιδιωτικούς πελάτες να δίνουν αυτήν την ε, δυνατότητα πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Γιατί το αφήνω αυτό στα κράτη-μέλη. Αυτό γιατί πρέπει να υπάρξει ισοδίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και δεν θα είχε νόημα οι τράπεζες που έχουν ιδιώτες ως πελάτες να πρέπει να παρέχουν λογαριασμούς και άλλες τράπεζες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό να μην υποχρεωμένες να δίνουν λογαριασμούς. Γι' αυτό προτιμώ να μείνει αυτό ανοιχτό στα κρατημέλη, ώστε τα κρατημέλη να εκτιμήσουν καλύτερα που υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού και που όχι. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη, όπως παραδείγματος στην Αυστρία, υπάρχουν συγκεκριμένες τράπεζες οι οποίες έχουν τέτοιου είδους λογαριασμούς μονάχα. Ερχόμαστε τώρα στα βασικά χαρακτηριστικά ενός βασικού τραπεζικού λογαριασμού και τι είδου συναλλαγές θα πρέπει να μπορούν να γίνουν με αυτό το λογαριασμό. Πιστεύω ότι όλες οι διαδικασίες για το άνοιγμα, το κλείσιμο και τη διαχείριση αυτού του λογαριασμού θα πρέπει να την χάνουν για τους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα σε ένα λογαριασμό και επίσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εντολές πληρωμής, μεταφορές πιστώσεων, αναλήψεις μέσα σε μια κάρτα ε, ε για, για να βγάζουν χρήματα από κάποιο μηχάνημα σε καθημερινό επίπεδο. Μια κάρτα αναλήψεων. Όλα αυτά λοιπόν ανήκουν στην καθημερινή λειτουργία ενός λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, να συνδέεται με την αγορά άλλων υπηρεσιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές λένε σε κάτι μέλη, ναι, ένας βασικός λογαριασμός, αλλά σας δίνουμε ένα βασικό λογαριασμό αν εσείς θα χρησιμοποιήσετε και άλλες υπηρεσίες της τραπεζάς μας, μια ασφαλιστική υπηρεσία ή οτιδήποτε τέτοιο. Όχι, ένας βασικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι ένας πρωτόγονος, απλός λογαριασμός, χωρίς καθόλου πρόσθετες υπηρεσίες. Θα πρέπει <clears throat> να εξασφαλίσουμε και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται προπληρωμένες κάρτες ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, οποιαδήποτε μορφή πιστοτικών καρτών χωρίς δικαίωμα να κάνει κανείς μια ανάληψη που ξεπερνάει τα χρήματα που βρίσκονται στον τραπεζικό λογαριασμό, του λεγόμενου overdraft. Να έχει δυνατότητα κανείς να έχει μια κάρτα όπως η πρώτον στο Βέλιο η οποία δίνει τη δυνατότητα μικροπληρωμών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιτρέπονται. Υπάρχουν σήμερα πολλοί λογαριασμοί βασικού χαρακτήρα που λειτουργούν μονάχα μέσα από το ίντερνετ. Αυτό μπορεί να είναι ιδανικό για ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά υπάρχει και ένα τμήμα του πληθυσμού που με τον τρόπο αυτό αποκλείεται. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι η μόνη δυνατότητα που θα δώσουμε μέσω του ίντερνετ άτομα τα οποία είναι άστεγα και δεν έχουν προφανώς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ηλικιωμένοι ή Καλά, οι φοιτητες φυσικά έχουν όλη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά μπορούν να είναι άτομα τώρα από τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα που για αυτά είναι πραγματικά δύσκολο να έχουν πρόσβαση από το διαδίκτυο σε ένα βασικό λογαριασμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτός ο απλός, ασφαλής και φιλικός προς το χρήστη για όλους τους πολίτες. Επίσης, όταν πρέπει να αλλάξει κανείς τράπεζα και εκεί πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να κάνει κανείς μια αλλαγή τράπεζα, και θα πρέπει στο βαθμό του δυνατού να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχει κόστος για αυτή την αλλαγή και αν πρέπει να καταβάλει κάποιο κόστος ο καταναλωτής θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι μόνο το διοικητικό κόστος που είναι απαραίτητο για την μεταφορά του λογαριασμού θα πρέπει να καταβάλλεται από τον καταναλωτή αλλά δεν πρέπει να του επιβάλλονται πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πρόστιμα ή τέλη εάν υπάρξουν καταστάσεις ανεξάτητη από την ε, θέληση του καταναλωτή, αν παραγωγός χάρη υπάρξει ακάλυπτο ποσό στο λογαριασμό του λόγω ε, καθυστέρησης καταβολής πληρωμών ή λόγω επιταγών οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί κτλ. Εγώ είχα αυτή την εμπειρία σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Είχα αλλάξει από εντολές προς την τραπεζά μου και παρόλα αυτά η τραπεζά μου πράγματι εξετέλεσε εντολές οι οποίες δεν καλυπτόντουσαν στο παρελθόν και ουσιαστικά κατέληξε σε μια διπλή πληρωμή από, την, από, το λογαριασμό αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι ανεξάρτητες της θέλησης του καταναλωτή δεν πρέπει φυσικά να υπάρχουν ε, πρόστιμα κατά του καταναλωτή. Αν υπάρξουν λοιπόν σύντομες, ε, σύντομα διαστήματα που είναι ακάλυπτος ο λογαριασμός, δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε πρόστιμα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία προβλέπουν μία μικρή δυνατότητα υπέρβαση στο λογαριασμό, ακόμα και στο βασικό λογαριασμό. Δεν ξέρω ποια κράτη-μέλη θέλουν να το διατηρήσουν αυτό το προνόμιο για τους καταναλωτές. Αν υπάρχει δυνατότητα λοιπόν μιας μικρής πίστοσης ακόμα και για το βασικό λογαριασμό σε ορισμένα κράτη-μέλη, κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να παραμείνει σε διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτή τη διευκόλυνση ή όχι. Στο βαθμό που αυτό φυσικά βρίσκεται σε λογικά πλαίσια. Τίθεται στη συνέχεια το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εγώ πιστεύω ότι τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή Θα πρέπει να διατηρήσουμε την προστασία αυτών των δεδομένων σε υψηλό επίπεδο και ιδίω για άτομα τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, παραγωγή χάρη σε κατάσταση ε, δεν θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα αυτών των ατόμων να τύχουν <clears throat> χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης, κάτι το οποίο θα θέσει σε αυτούς τους καταναλωτές σε μια δύσκολη κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δίνουμε σε αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση. Επίσης, το, το δικαίωμα προσφυγής και η υποβολή παραπώνων υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις τράπεζες, αλλά σε άλλα κράτη-μέλη δεν υπάρχει μηχανισμός για την αντιμετώπιση των παραπώνων και των προσφυγών Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα πρόσθετο μηχανισμό για την επίλυση διαφορών και παραπώνων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι βασικές προδιαγραφές. Η υπερβολική πολυμορφία εδώ πέρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες τους. Όταν μιλάμε επίσης για ε, διαφάνεια και για πληροφόρηση σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών και αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι είναι φιλική προς τον ε, χρήστη οι πληροφόρηση που έχουν σε σχέση με τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο βασικός λογαριασμός. Για την εφαρμογή και την εποπτεία αυτού του, αυτής της οδηγίας. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέχρι δύο χρόνια μετά την θέση εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας να μας δώσει μια πλήρη έκθεση για την εφαρμογή και την λειτουργία αυτής της οδηγίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορούμε, αν προκύψουν προβλήματα, το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε αυτή την οδηγία, πάντα φυσικά προς την κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών μακρηγόρησα σήμερα γιατί θεώρησα ότι ήταν χρήσιμο να σας παρουσιάσω την πλήρη παλέτα των θεμάτων που συνάπτονται με αυτή την οδηγία και είχα βέβαια και την πρώτη επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές είχα επιπλέον επαφές με τον εισηγητή της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και η άποψή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε δυνατότητα να έχουμε μια ευρεία συνένεση για τα θέματα αυτά και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία τους και για όλες τις προτάσεις οι οποίες έχουν βελτιώσει την έκθεσή μου. Θα καταθέσω και εγώ ίδια κάποιες τροπολογίες, γιατί δεν μπορούσα να καλύψω όλα αυτά τα οποία ήθελα να αναφέρω λόγω του περιορισμού στο μήκος μιας έκθεσης, αλλά σίγουρα με τροπολογίες νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω αυτά τα οποία θα ήθελα να βάλω στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε, Εύλην για την υποστήριξη που δώσατε σε αυτή τη σημαντική πρόταση και την ευσυνειδησία με την οποία έχετε φέρει σε πέρα στο έργο σας. Και εγώ είμαι απογοητευμένος που δεν μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ισότιμη σχέση με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, αλλά έχουμε προωθήσει αρκετά το θέμα αυτό και με την ακρόαση και νομίζω ότι θα επηρεάσουμε σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω λοιπόν θα έχουμε την επιρροή που θέλουμε. Έρχομαι στους κοιόδες εισηγητές. Πρώτος είναι ο Hans Peter Μάιερ και όποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Hans Peter Μάιερ, Schmidt, Τούρουνεν κτλ. Σας ευχαριστώ λέει κύριος Μάιερ, Hans Peter Μάιερ. Θέλω να αναγνωρίσω το σημαντικό έργο της κυρίας ε, Gebhardt και για τη συστηματική αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων στην έκθεσή της. Δεν έχω πολλές τροπολογίες, γενικά υποστηρίζω απόλυτα το έργο της εισηγήτριας. Ίσως μια προσθήκη, κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί περισσότερο, ότι πρέπει η πρόσβαση στο βασικό λογαριασμό να γίνεται χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, ώστε κάποιο ο οποίο παραδείγματο χάρη θέλει να κάνει μια σύμβαση μίσθωση να έχει αυτό το λογαριασμό, αλλά να μην συνδέεται ο λογαριασμό αυτό με άλλε υπηρεσίε οι οποίε θα του επιβληθούν. Ή παραδείγματο χάρη να πρέπει να παρουσιάσει την, ε, την, ε, το συμβόλαιο μίσθωση για να μπορεί να έχει τον βασικό λογαριασμό ο καταναλωτή. Τώρα για τα θέματα δικαιοδοσίας θα θέλω να είμαι πιο σαφής και συγκεκριμένος. Έχουμε δει ότι η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων θα είναι η επιτησή της αρμόδια. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση ώστε να ληφθούν υπόψη και οι αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. <clears throat> Νομίζω ότι έχουμε μια καλή συμβιβαστική πρόταση που καταθέσαμε. Τελικά είναι λιγότερα αυτά τα οποία επιτύχαμε και αυτό με στενοχωρεί. Δεν, με, δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο έγινε. Αυτό το οποίο από την άλλη πλευρά είναι θετικό είναι ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ χθε και ενώπιον των δημοσιογράφων έκανε σημαντικές δηλώσεις γιατί είπε ότι ακόμα και για τους κανονικούς λογαριασμούς είναι απαραίτητη να υπάρχει διαφάνεια <clears throat> για τα τέλη τα οποία επιβάλλονται για τραπεζικές συναλλαγές. Ότι δεν είναι κάτι το δεδομένο λοιπόν στη σημερινή στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε και νομοθεσία η οποία να λέει με σαφή τρόπο ότι πρέπει να υπάρχουν νομικοί κανόνες, νομικής ισχύω κανόνες, όπως λέει και ο κύριος Μπαρνιέ, που θα εξασφαλίσουν ότι ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε αυτό το βασικό λογαριασμό. Στο παρελθόν η Κομισιόν και ο κύριος Μπαρνιέ βασιστήκαν στην αυτορύθμιση, ήλπισαν ότι αυτό θα λειτουργήσει, αλλά αυτό δεν έχει λειτουργήσει. Επομένως θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε ότι η Κομισιόν θα προχωρήσει και θα θέσει και μια νομοθετική πρόταση με το περιεχόμενο το οποίο έχουμε συζητήσει. Θα πρέπει όμως παράλληλα και η Κομισιόν να μας πει ποιο είναι το κεντρικό σημείο της πρότασής της. Θα είναι μια πρόταση για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα ή θα είναι αυτό το οποίο ζητούμε εμείς μια πράξη για την προστασία των καταναλωτών. Για μένα αυτό το θέμα αφορά την, προστασία των ε, πολιτών έναντι των τραπεζών. Και από εκεί έλκεται η επιτυσίλης αρμοδιότητα οι τράπεζες φυσικά εμπλέκονται, αλλά οι τράπεζες καλούνται να υλοποιήσουν ένα δικαίωμα των πολιτών, όχι μια υποχρέωση των πολιτών. Επομένως εμείς ως Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών, εμείς θα έπρεπε να έχουμε την θέση της καθήλυνα αρμόδιας Επιτροπής. Επομένως, αν η Κομισιόν είχε διατυπώσει σαφέστερα την πρότασή της, θα ήταν πιο εύκολο να ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες και στο Κοινοβούλιο, γιατί θα ξέραμε ποιος θα ήταν αρμόδιος επί της ουσίας. Αλλά τονίζω και πάλι ότι θέλουμε να εργαστούμε για μια νομοθετική λύση για το θέμα αυτό. Δεύτερον, να πούμε ότι είναι μια νομοθεσία η οποία ασχολείται με τα δικαιώματα και την απέτηση των καταναλωτών να έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό και η κύρια μέρημνα τη ε, πρόταση τη Κομισιόν εμείς πρέπει να είναι η προστασία των καταναλωτών και όχι η ρύθμιση των τραπεζών. Κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Γκέπχαρτ. Νομίζω ότι είναι άκρας σημασία η έκθεση αυτή. Εγώ είμαι υπέρ της αυτορύθμισης. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδου εργαλεία πότε πότε. Όμως, στην περίπτωση αυτή, μάλλον το πράγμα διαφέρει λίγο. Μιλούμε για τράπεζες που είναι μέρος της ε, κοινωνίας, του κοινωνικού συστήματος. Ξέρουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων <clears throat> επέτρεψαν να διασωθούν πολλές τράπεζες ανά τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και εμείς το επιτρέψαμε αυτό. Οι υπουργοί το επέτρεψαν, διότι είναι ένα ζωτικό τμήμα του όλου συστήματος πληρωμών. Με αυτό το είδος τα επιχειρήματα λοιπόν και τα προηγούμενα, μπορώ και εγώ ίδιος να δεχτώ ότι πραγματικά μιλάμε εδώ για ένα βασικό δικαίωμα των πολιτών. Ακόμα και αν πιστεύω λοιπόν στην αυτορύθμιση, τι να καταλήγω να μην έχω αντίρρηση. Παρόλο που είμαι επί της ουσίας ε, φιλελεύθερος και φιλελευθεριστής. Αλλά το πρώτο ερώτημα είναι πιστεύει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπαρνιέ ότι μπορεί να ετοιμαστεί νομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό, γιατί ένα χρόνο πριν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Περίεργο λοιπόν. Όμω, καλό θα ήταν να επηρεαστεί αυτό το σύστημα. Το χρειαζόμαστε και υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου βασιλεύει το χρήμα, το μετρητό. Εάν θέλουμε να είναι ασφαλέστερη η κοινωνία μας, η χρήση πιστοτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών, θα πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως και να το σχεδιάσουμε αυτό. Ίσως μέτρα για την αντιμετώπιση της λεύκανσης ε, χρήματος προσόδων ή για την παραποίηση, ίσως αυτά να μπορούσαν να συνδυαστούν εδώ. Είμαι λοιπόν, την να υπέρ της πρότασης. Αλλά θα ήθελα να σταθώ και σε κάποια σημεία. Ε, I think ε, there at least five. Τουλάχιστον πέντε. Πρώτα απ' όλα, ισορροπία και το κόστος για τους καταναλωτές και τους παρέχοντες. Έπειτα η διασφάλιση πραγματικής επιλογής και εναλλακτικών για τους καταναλωτές με ευρύ φάσμα παρεχόντων αυτές τις υπηρεσίες. Έπειτα ένας επαρκής μηχανισμός επίλυσης προσφυγών. Τέταρτο, να συμφωνήσουμε τι είναι, ποιος είναι ο ορισμός και το τι εμπεριέχει ο ορισμός του βασικού λογαριασμού κάρτα πληρωμών λόγου χάρη θα συμπεριλαμβάνει. Και πέμπτον, να δούμε πώς θα διευκολύνουμε την κινητικότητα για όλους τους νομικούς κατοίκους, τους νόμιμους κατοίκους μάλλον. Αυτό <clears throat> το συμφωνήσαμε και στην ε, συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Θα πρέπει να δούμε τι θα σημαίνει η νόμιμη κατοικία και τι τεκμηρίωση θα απαιτείται. Τι παραστατικά. Λοιπόν, νομίζω Το βασικό επιχείρημα και η βασική πρόταση θα πρέπει να ακουστεί από την Επιτροπή μα. Και εδώ είμαι αναπληρωτή, αυτό πρέπει να το πω. Ε, θέλω να μιλήσω από τη διπλή ιδιότητα λοιπόν του αναπληρωτικού μέλου εδώ και αναπληρωματικού μέλου εδώ και πλήρου μέλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, ε, έκφραση όλων αυτών σε νομική πρόταση. Για μια σειρά από λόγους, οικονομικούς, λόγους υπέρ των καταναλωτών, χρειαζόμαστε αυτή την πρόταση για τα νόμιμα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω λοιπόν να το πετύχουμε και να έχουμε μια καλή συμβαστική πρόταση που να προέλθει και από τις δύο επιτροπές. Πρόεδρο, ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Κυρία Τουρούνεν. Ευχαριστώ. Ως προς τις αρμοδιότητες, και εγώ συμμετέχω και στις δύο επιτροπές και επί της ουσίας στην ίδια λογική βρισκόμαστε. Είναι παρόμοιες οι δύο εκθέσεις, δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Επί της ουσίας, ωραία, θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει υπέρ της ε, έμφαση θα πρέπει να δώσουμε στα τραπεζικά ζητήματα εδώ. Οι τράπεζε θέλουν κάποιε υπηρεσίε να συμπεριλαμβάνονται. Κάποιο άλλο υπέρ τη ε, διάθεση των καταναλωτών. Θα μπορούσαν να υπάρξουν διαφωνίε, θα μπορούσα και εγώ να επιμείνω, αλλά όπω είπε και ο κύριο Σμιτ, εκτό κοινοβουλίου αυτό που ζητούν οι άλλοι από εμά είναι ένα σαφέ αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω που να επιδιώξουμε. Επί το περιεχομένου καλωσορίζουμε την έκθεση, συμφωνούμε με όλα τα βασικά σας επιχειρήματα και οι προτεραιότητές μας καλύπτονται. Ναι, όντως πρώτον χρειαζόμαστε μια οδηγία, δεύτερον θα πρέπει να δηλώσουμε με σαφήνεια ότι μιλάμε εδώ για δικαίωμα των καταναλωτών και καθήκον του να επιτρέπονται αυτέ οι πληρωμέ. Τρίτον, ότι θα πρέπει να είναι εύκολη πρόσβαση στο δικαίωμα αυτό. Και τέταρτον, ότι θα πρέπει να δώσουμε λεπτομερέστερη περιγραφή των χαρακτηριστικών. Τι είναι ο βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό το επιχειρήσατε και συμπεριλαμβάνεται σε ένα βαθμό. Και πέμπτον, χρειάζονται πληροφορίε για να είμαστε βέβαιοι ότι όχι μόνο στην νομοθεσία μας θα συμπεριληφθεί αυτό το μέτρο, αλλά θα το κατανοήσουν και οι πολίτε. Θα ξέρουν τι εννοούμε. Νομίζω λοιπόν ότι λίγο πολύ συμφωνούμε. Απλώς από τους πράσινους θα θέλαμε κάποιες περισσότερες ε, λεπτομέρειες στη διατύπωση, να είμαστε ακριβέστεροι για τις πληρωμές λόγου χάρη, τι θα κοστίζει. Δίκιο έχετε όταν λέτε ότι θα πρέπει να είναι ή δωρεάν ή σε εύλογο κόστος, ίσως απλώς να το εξηγήσουμε αυτό, να μην υπερβαίνει λόγου χάρη το κόστος παροχής της υπηρεσίας κτλ. Επίσης, για το ποιες τράπεζες αφορά αυτό. Θα μπορούσε να το αναλάβει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων βέβαια, αλλά και εδώ χρειάζεται ακριβέστερη διατύπωση. Ποιες ακριβώς τράπεζες υποχρεούνται ή θα υποχρεούνται να προσφέρουν πρόσβαση σε τέτοιο λογαριασμό και ποιες όχι. Μπορεί ας πούμε οι κεντρικές τράπεζες ε, θα μπορούσαν, σε καμία περίπτωση βέβαια, ή άλλοι, τέλος πάντων μικρές τράπεζες, θα δούμε, θα το σκεφτούμε. Επίσης το θέμα της επίλυσης διαφορών και εκεί να γίνουμε κάπως αφέστεροι στη διατύπωση, να το διασυνδέσουμε με κάποιους υπάρχοντες ήδη μηχανισμούς, να μην επινοήσουμε νέους, λογικό είναι αυτό, συμφωνούμε, και κάποιες τροπολογίες θα υποβληθούν για να κάνουμε κάποιες προσθήκες σε όσα ήδη μας εξηγήσατε. Επίσης, κάτι για το οποίο δεν έχω αποφασίσει είναι η δυνατότητα υπερχρέωσης δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό εφόσον ανοίγουμε ένα βασικό λογαριασμό από τη μία να προβλέπουμε τέτοια δυνατότητα. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να το συζητήσουμε. Για παράδειγμα, μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό περιθώριο υπερχρέωση. Να το συζητήσουμε λίγο, γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε από τώρα. Εντάξει, δύσκολο. Τίνω να σκεφτώ ότι μπορεί να μην είναι πολύ ρεαλιστικό να μείνουμε στο ασφαλές πλαίσιο ότι εντάξει, ας πάρουμε το λογαριασμό που μπορεί όλοι να δεχτούν και τα, να τα αφήσουμε, αλλά ας είμαστε ανοιχτοί σε μια πρώτη συζήτηση. Εγώ προσωπικά δεν έχω αποφασίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο λόγια και από μένα για εξ ονόματος του σκιώδους της ομάδας μου που είμαι εγώ. Μπορεί να μείνουμε εδώ αύριο, αλλά θέλω να πω ότι η θέση του είναι πολύ κοντά στο κυρίου Σμιτ. Εμείς δεν έχουμε άποψη βασικά. Θα δούμε τι θα γίνει στη συζήτηση, αλλά χαίρομαι που η κυρία Γκέμπχαρτ συμπεριέλαβε το θέμα ότι μπορεί να μην είναι αναγκαστικά τράπεζες που θα χορηγούν αυτή την υπηρεσία στους χρήστες των κινητών. Αλλά πράγματα όπως οι προπληρωμένες κάρτες κλπ. Ήταν πρόταση που πολλοί έφεραν, τις έφεραν αντιρρήσεις. αλλά κοινωνίες που έχουν μικρή πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς θα μπορούσαν να υποφεληθούν. Επίσης τα εμβάσματα είναι χρήσιμα γιατί πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν αυτές τις προπληρωμένες κάρτες που έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες σε πολίτες που δεν είχαν πρόσβαση σε τράπεζες. Χρησιμοποιούν μια προπληρωμένη κάρτα και έτσι κινούν το κινητό τους. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι αν υπάρξει τέτοιο νομικό πλαίσιο να μην περιορίζεται στις τράπεζες. Μπορεί να θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση προμηθευτών και υπηρεσιών πέραν των τραπεζών, οι οποίες είναι σε τέτοια πίεση τώρα με την κρίση για να χορηγήσουν δάνεια που αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους, παραδείγματος χάρη δεν δανείζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως πριν. Και το μέλλον πολλών από αυτές είναι αβέβαιο. Ίσως και άλλες καινοτόμες μέθοδοι όπως οι προπληρωμένες κάρτες να είναι μια λύση. Να το σκεφτούμε λοιπόν με πιο ευρύ πνεύμα, όχι μόνο τις τράπεζες ως προμηθευτές πρόσβασης σε μηχανισμούς πληρωμής. Θα τα πούμε όλα αυτά και στη συνεδρίαση των σκιωδών. Θέλει κανείς άλλος, ο κύριος Διόν, είστε και εσείς σκιώδης, α, σας ξέχα ξεχάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω εδώ ένα προβληματάκι γιατί εγώ βλέπω τα πράγματα ως θέμα πρωτοβουλίας καταναλωτών και καταναλωτριών. Από την άλλη, συνεννοήθηκα και με άλλους κοιόδης και ίσως να πρέπει τις ιδέες της κυρίας Γκέπχαρτ όντως να τις συμπεριλάβουμε και εμείς. εγώ και η ομάδα μου εγκρίνουμε την έκθεση της κυρίας Γκέπχαρτ και δεν έχουμε πολλά να σχολιάσουμε από αυτής. Ίσως στη σύσταση 2 όπου αναφέρεται η υποχρέωση των τραπεζών να διασφαλίζουν τις βασικές πληρωμές αλλά επίσης να δικαιολογούν την τυχόν αρνήσεις. Ίσως εδώ πρέπει να μπει και κάτι άλλο μεταξύ των δύο. Ότι δεν μπορούν να αρνούνται παρά μόνο με σοβαρούς λόγους κτλ. Δεν συμφωνώ όμως τελείως με αυτά που είπε ο πρόεδρος για τα κινητά. Διότι νομίζω ότι ένας τραπεζικός λογαριασμός προσφέρει πολλά περισσότερα από ότι μία προπληρωμένη κάρτα ή κάρτα προπληρωμής. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ποσά από το κινητό. Ούτε μπορεί η προπληρωμένη κάρτα να έχει όλες τις χρήσεις του κανονικού λογαριασμού. Εγώ μένω στις ιδέες της κυρίας Γκέμπχαρτ Ναι, συγγνώμη που σας είχα ξεχάσει. Λοιπόν, μίλησαν όλοι οι σκιώδεις. Ίσως προλαβαίνει τώρα και η Κομισιόν να σχολιάσει και μετά ξανά η κυρία Γκέμπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης για την προετοιμασία της λεγόμενης δέσμης των τραπεζικών λογαριασμών. Σήμερα αρχίζει η δημόσια διαβούλευση για το κόστος των τραπεζικών υπηρεσιών. Είχε γίνει μια προσπάθεια αυτορύθμισης αλλά δεν πέτυχε και υπάρχει και το θέμα του account switching που είπε και η κυρία Γκέμπχαρτ. η Κομισιόν έκανε μερικές έρευνες για το λεγόμενο mystery shopping. Έτσι για να δούμε αν όντως δουλεύει πρέπει να το ξαναδούμε και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. οι πληρωμές για όλους τους ε, ιδιοκτήτες ή χρήστες τραπεζικών λογαριασμών είναι κάτι που θα το εξετάσουμε η ασφάλιση των πληρωμών. Και όποιοι έχουν ιδέες μέχρι τέλη Ιανουαρίου να μας τις πούν. Ακόμη όμως περιμένουμε απαντήσεις. Αν θέλετε κύριε Πρόεδρε να μιλήσει και η συνάδελφός μου εδώ για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα στις χώρες μέλη. Καλημέρα σας. Μέχρι σήμερα λάβαμε 20 προτάσεις από 6 χώρες μέλη τα 14, α, 14 άλλα κράτη-μέλη επέλεξαν να μην κάνουν τίποτε, να μην αντιδράσουν προς τη σύσταση και τα περισσότερα από αυτά τα κράτη δεν προβλέπουν κανένα ειδικό νομικό πλαίσιο για αυτό το θέμα. Μάλιστα σύντομα. Όσο για το σχέδιο πρωτοβουλίας λέει ο μιλητής, γνωμοδότησης δηλαδή, θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Βεβαίως δεν είναι ταυτόσιμο με τις προτάσεις μας, αλλά δικαίωμά σας είναι. Παίρνουμε υπόψη μας πάντως όλα όσα ακούστηκαν εδώ για τις λεγόμενες λιανικές τράπεζες. Το θέμα της ενδιάμεσης ζώνης που ανέφερε η κυρία Γκέμπχαρτ είναι πρόβλημα που υπάρχει μόνο σε μερικές χώρες μέλη όπως τη Δανία. Η, το δικαίωμα σε μια διευκόλυνση overdraft ε, είναι ευαίσθητο θέμα, συζητιέται όμως και για τις προπληρωμένες κάρτες είναι κάτι που το βρίσκουμε ενδιαφέρον αν και δεν το προβλέπει η σύσταση. Όπως σας είπα όμως ακόμα είμαστε σε διαβούλευση και οποιαδήποτε καλή ιδέα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την κυρία Γκέμπχαρντ ιδέες και από όλους τους κοιόδες. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκέμχαρντ, αν θέλετε να συνοψίσετε, έχουμε κανένα λεπτό περίπου. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο είμαστε στον σωστό δρόμο. Και όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε μια εκθέση νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να παροτρύνουμε και να βοηθήσουμε την Κομισιό να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και εγώ θα ήθελα ο κύριος Πάρκε και η Κομισιό να είχαν προχωρήσει σε ένα νομοθέτημα, σε μια πρόταση νομοθετήματος γιατί αυτό προεβλέπεται στο νομοθετικό της πρόγραμμα για το 2011. Ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα βέβαια, πολλές φορές γίνεται μία πρόταση, αλλά είναι πολλές φορές δύσκολα στα νομοθετικά κείμενα να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Πολλές φορές ξεχνάνε τις διστάσεις. Ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι για όλα αυτά που είπατε και πάλι γιατί πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα απόρριψης αυτού του δικαιώματος από τις τράπεζες. Δεν έχω ίσως αναφερθεί σε σχέση με αυτό το θέμα επαρκώς στην εκθεσή μου. Πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο, αλλά απλώς να επισημάνω το ότι υπάρχει περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις ε, ξεπλήματος χρημάτων ε, και διαφθοράς που θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Θα πρέπει να αφήσουμε στις τράπεζες τη δυνατότητα να κάνουν μια εξαίρεση του δικαιώματος που προβλέπεται από την έκθεση αυτή και να μην ανοίξουν λογαριασμό σε ορισμένα άτομα. Αλλά φυσικά αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε μια σαφέστερη διατύπωση για να είναι σαφές με τι είδους επιχειρηματολογία μπορεί μια τράπεζα να αρνηθεί να ανοίξει αυτό το βασικό τρόπο λογαριασμό και φυσικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου διατάξεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τρόπο, ε, λογαριασμό και το χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα αυτού του λογαριασμού. <clears throat> Μπορούμε ίσως να αλλάξουμε την ε, διατύπωση εδώ. Τώρα, σε σχέση με τη χρήση τηλεφώνων για την διακίνηση λογαριασμών, αυτό υπάρχει όπως ξέρετε και εξελίσσεται όλο και περισσότερο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν προτείνει αυτό σαν μια αναλλακτική μορφή λογαριασμού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτό να συνδέεται με την ύπαρξη ενός πραγματικού και όχι μονάχα εικονικού λογαριασμού. Να έχουμε διαχείριση με το τηλέφωνο, αλλά πρέπει κάπου η τράπεζα να κρατάει τα πραγματικά χρήματα. Τον βασικό αυτό λογαριασμό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα υπάρχει πάντα ανεξάρτητα από τη διακίνηση από τηλέφωνο ή όχι. Και αγαπητέ Μάλκομ, εκεί συμφωνώ μαζί σας. Αλλά νομίζω είναι μια καλή δυνατότητα, αλλά δεν είναι επαρκές μόνο με το τηλέφωνο να γίνει τη διακίνηση του λογαριασμού. Να έχει κανείς ένα λογαριασμό από το τηλέφωνο δηλαδή. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένας πραγματικός λογαριασμός που είναι αυτός ο βασικός λογαριασμός. Δεν έχω τώρα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτή την έκθεση γιατί δεν ήταν σαφές για μένα αν μέσω της ε, <clears throat> απόφασης της συνέλευσης των Προέδρων θα εξακολουθήσει να είναι έγκυρο το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Βλέπω ότι τώρα η γραμματεία σας ε, δίνει κάποια στοιχεία και επομένως θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας θέση στο σημείο αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθούν οι διαπραγματεύσει σα με την ε, οικονομική. Συνεχίζουν οι διαπραγματεύσει με την Οικονομική και, και Νομισματική Επιτροπή. Νομίζω ότι προβλέπουν να ψηφίσουν στις 29 Μαΐου για τα θέματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε τα χρονοδιαγράμματα, αλλά προς το παρόν η προθεσμία τροπολογία τροπολογιών για την εκθεσή σου έβλενε στις 3 Απριλίου το μεσημέρι. Θα τις εξετάσουμε στις 8 Μαΐου και θα ψηφίσουμε στις 29 Μαΐου. Βέβαια θα πρέπει τότε η Οικονομική Επιτροπή να προσαρμοστεί σε εμά, αφού δεν θα έχουμε συνεδρία στις ψηφοφορία. Και θα πρέπει να υπάρχει χρόνος διαπραγματεύσεων για να συμπεριληφθούν δικές μας τροπολογίες στην έκθεσή τους. Το σημαντικό είναι προθεσμία για τροπολογίες 3η Απριλίου το μεσημέρι. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε στο σημείο αυτό. θα ήθελα, αν με ακούει, να εξάρω και τη συμβολή σε αυτή την έκθεση της κυρίας Μπαρνεμαρτίνες, η οποία έχει εργαστεί ιδιαίτερα για την έκθεση αυτή. Είναι τελευταία της ε, παρουσία ως μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής μας, γιατί θα πάει σε μια νέα μονάδα με ένα προϊστάμενο ο οποίο ήταν παλιό υπαλληλό μας για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Λυπούμεθα που θα φύγει, αλλά θα παίξει και σε αυτή τη νέα μορφή, σε αυτή τη νέα μονάδα. Ε, <clears throat> καλή τύχη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μπλάνκα για την βοήθειά σου στην Επιτροπή μας. Ένα θέμα special τώρα. Ο καθηγητής Κρέν βρίσκεται κάτω στα θεωρία, αλλά στη, στα έδρανα των ε, παρισταμένων, αλλά ίσως ε, θα ήθελε να έρθει εδώ πάνω. Αλλά θα δώσετε την ε, παρουσίαση, μήπως εμείς να κατέβουμε κάτω. Να σας παρουσιάσω λοιπόν από τα υψίπεδα στα οποία βρισκόμαστε. Έχετε επεξεργαστεί μια πολύ σημαντική έκθεση για τις τεχνολογίες που δημιουργούν ικανότητες. Τις ικανοποιητικές επομένως τεχνολογίες. Αυτό γι' αυτό ενδιαφέρεται όλη μας η Επιτροπή και φυσικά έχετε παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκθεση της ομάδος εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Ξέρω ότι για κάθε μεγάλο σοφό υπάρχουν πάντα και οι Σέρπα οι οποίοι κάνουν την ούτως υπήν γαϊδουροδουλειά της έκθεσης αυτής. Ο ρόλος της ομάδας Σέρπα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο καθηγητής Κριν ήταν ο πρώτος της ομάδας των ε, Σέρπα, επομένως ξέρει καλύτερα από τους άλλους ποια είναι τα θέματα αυτά. είναι ε, διευθυντής της Επιστημονικής Επιτροπής της Γαλλικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Υπήρξε, βλέπω τώρα εδώ πέρα ένα μακρινάρι στο βιογραφικό του, ίσως θα μας πει αυτός περισσότερα. Είναι τόσο μακρύ το βιογραφικό του που δεν έχω προλάβει να το διαβάσω και εγώ. Θα του δώσω όμως αμέσως το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση αντίγραφα της ε, παρουσίασης και μετά θα υπάρξουν ερωτήσεις. Εγώ κατεβαίνω για να δω καλύτερα τις διαφάνειες. Ε, thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση ώστε να κάνω αυτή την παρουσίαση σήμερα. Η παρουσίαση αυτή δεν αφορά την τεχνολογία, αφορά τις θέσεις εργασίας. Και οι Financial Times έλεγαν ότι 10,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι σήμερα το πρωί. Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή λοιπόν θα μας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποια τα ζητήματα που σήμερα μας απασχολούν. Να τα πω γρήγορα. Τέσσερα βασικά μηνύματα από την έκθεση θέλω να σας ε, εντυπωθούν. Πρώτα απ' όλα ότι οι κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, ΚΤΕ, είναι καθοριστικές για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Καταλαβαίνω ότι αυτό αναγνωρίστηκε και συνόδο του Συμβουλίου πριν από λίγες εβδομάδες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνθηκε να εντείνει τις δραστηριότητά τη σε σχέση με τις ΚΤΕ. Έπειτα, η Ευρώπη είναι άριστη στα επιστημονικά ζητήματα, αλλά δεν μπορεί να την ε, μετατρέψει σε προϊόν την επιστήμη στην παγκόσμια εργονά. Και έχουμε πρόβλημα με το μερίδιο αγορά παγκοσμίω και τι θέσει εργασία που δημιουργούμε. Το επόμενο μήνυμα είναι ότι πρέπει να δούμε προσεκτικά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία άλλαξε το όνομα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας σε Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας. Η προσθήκη όμως ενός όρου, η προσθήκη όρου στον τίτλο μιας Γενικής Διεύθυνσης δεν αλλάζει κατά την ουσία. Θα πρέπει να ενισχυθεί ως ο ανάλογος προπολογισμό. Τέλο, ελπίζω θα μπορέσετε και εσεί να παροτρύνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα έχουμε εντατικέ σχέσει συνεργασία μεταξύ των κονδυλίων για την καινοτομία και τα διαφορετικά κονδύλια και την ανάπτυξη των ΚΤΕ. Θα είμαι σύντομο και στο τέλο θα σα αφήσω χρόνο και για ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, οι ΚΤΕ εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 για κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, για την γνώση, για το υψηλό ποσοστό δυναμικού που επιτρέπουν και για την ε, συσχετισμό τους με την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν έγιναν κάποιες συστάσεις για τις ΚΤΕ και η ομάδα υψηλού παρέμεινε σε έξι βασικές. Η σημασία των ε, ΚΤΕ είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν με συγκεκριμένα προϊόντα σήμερα. Ας δούμε ένα ηλεκτρικό όχημα του μέλλοντος με προηγμένα συστατικά, όπως την μπαταρία του αυτοκινήτου. Χρειάζονται ηλεκτρονικά για το τιμόνι, για τα παράθυρα. Χρειάζεται γνώση ε, ηλεκτρική για τα φώτα του αυτοκινήτου, για τα λάστιχα του αυτοκινήτου, νανοτεχνολογικές γνώσεις, για την βαφή του αυτοκινήτου, λόγου χάρη, και συνολικά για την κατασκευή τεχνολογικά μέσα. Η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί στην, ε, σε ηγετικό ρόλο για τις ΚΤΕ. Αλλά είτε μιλάμε για ηλεκτρικό όχημα είτε για κινητό τηλέφωνο, αυτό που βλέπουμε με αυτά τα κύρια προϊόντα, βλέπουμε ένα συνδυασμό πλέον τεχνολογικών μέσων. Δεν αρκεί μία από τις ΚΤΕ ε, για τα ηλεκτρονικά λόγω χάρη τα φωτοελεκτρικά, όχι. Είναι πολλές μαζί. Αν δούμε το iPhone της Apple, μια από τις ε, πιο πλούσιες εταιρείες των κόσμο. Έχει το γυαλί μπροστά, έχει πίσω την χρήση φωτοηλεκτρονικών στοιχείων. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται. Η τέταρτη πρόκληση που εντοπίσαμε στην έκθεσή μας είναι ότι αν χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό των ΚΤΕ, δυστυχώς, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πράξουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει χωρίσει σε διαφορετικέ γενικέ ε, διευθύνσει. Τα ηλεκτρονικά και τα φωτοελεκτρονικά είναι σε μία γενική διεύθυνση, τα υλικά και οι κατασκευέ στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα, και κάποια βιοτεχνολογικά προϊόντα σε άλλες ε, γενικές διευθύνσεις. Λοιπόν, ε, πρέπει να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την προώθηση των ε, Δεν είναι όμως μόνο σημαντικό να αναπτυχθούν αυτές τι τεχνολογίες, αλλά και να εξαπλωθούν, να διαδοθούν. Βλέπουμε ένα σημαντικό προϊόν σήμερα, ένα πλαστικό σωλήνα, οι οποίοι μπορεί σήμερα να μεταφέρουν καλώδια, νερό και όπως ξέρετε σε αστικά κέντρα, όταν κανείς κάψει στους δρόμους, Πολλέ φορέ μπορεί να σπάσει και έναν αγωγό, ένα σωλήνα, οπότε να διακοπούν επικοινωνίε ή ροέ. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ είναι να υπάρχει ένα σήμα, με ένας πομπός ε, στο σωλήνα. Αυτό είναι επαναστατικό για ένα τέτοιο προϊόν και ανοίγονται νέες αγορές για την Ευρώπη. Είναι τελείως νέο προϊόν. Μπορούμε λοιπόν τη ΚΤΕ να τις εισάγουμε και σε απολύτως παραδοσιακά προϊόντα. Εάν δούμε τις ε, βασικές αλυσίδε αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι είτε μιλάμε για αυτοκινητοβιομηχανία, είτε για τα φωτοελεκτρονικά, είτε για είναι ηλεκτρονικά, ΚΤΕ μπορούν να επηρεάσουν όλε αυτέ τι αλυσίδε. Εάν χάσουμε όμω τι ΚΤΕ, χάνουμε και την αλυσίδα αξία, όπω έχει ονομαστεί, και κάτι που έχει γίνει επανειλημμένο. Είναι λοιπόν στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, Εάν δούμε τώρα τι κύριε τεχνολογίε ευρύ εφαρμογή στην κατασκευή λόγου χάρη, ένα παράδειγμα, μια μικρή πόλη τη Άλπη, όπου έχουν ήδη κάποιους εξοπλισμούς, αλλά εάν δούμε τον όλο κατασκευαστικό τομέα, 5.000 θέσεις εργασίας απασχολούνται εδώ, αλλά 100 επιχειρήσεις γενικότερα. Δηλαδή υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με παρόχους, με διαμέσους, με λιανοπολιτές. Και αν δει κανεί το σύνολο της αλυσίδα αξίας, η κατασκευαστική αυτή μονάδα έχει να ε, να απασχολείται και να έρχεται σε επαφή με 300 μικρομεσαίες σε όλη την Ευρώπη. Εάν χαθεί λοιπόν αυτό, χάνεται όλο αυτό το δυναμικό καινοτομία. Όλε αυτέ οι δυνατότητε. Και αυτό δυστυχώ συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η κατασκευή και ο κατασκευαστικό τομέα δεν ακολουθεί την έρευνα. Η έρευνα ακολουθεί τον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό το βλέπουμε επανειλημμένω να συμβαίνει. Προχωρώντα τώρα, το δεύτερο μήνυμά μου αφορά τα επιστημονικά μα προϊόντα, την παγκόσμια αγορά και το μερίδιό μα και την απασχόληση. Κάποια στατιστικά στοιχεία. Αυτά τα ετοιμάσαμε για του επιτρόπου μα και προσπαθήσαμε να είναι απλούστατα για να τα καταλαβαίνουν. Το τρίγωνο δείχνει το μερίδιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνία που κατέχουμε σε τρει βασικέ ζώνε. Ε, Ευρώπη, Ηνωμένε Πολιτείε, Ασία. Αν δούμε τι ηλεκτρικέ μπαταρίε λόγου χάρη, θα θα δείτε ότι έχουμε 31% των διπλωμάτων στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε 30% και η Ασία 87%. 35% συγγνώμη. Ίσως έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων. Όμως εδώ το πλεόνασμα έρχεται από την ε, κατασκευή και από τη δημιουργία θέσεων εργασία. <clears throat> Δεν έχουμε τόσε πολλέ δυνατότητε για τα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χάρη. Ε, ε, χρηματοδοτούμε την επιστήμη, χρηματοδοτούμε και την έρευνα υλικών, αλλά δεν έχουμε αρκετή κατασκευαστικό τομέα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν 1% το 2008, διότι πολύ γρήγορα αργά περνάνε τα στοιχεία για τα διπλώματα μέσα από το σύστημα. Αλλά σήμερα πού επικεντρωνόμαστε σε ομοσπονδιακό και ε, επίπεδο από τις Ηνωμένε Πολιτείε σε δράσεις για να προσελκύσουν ξένες ε, εταιρείε με πρωτότυπα για τι ηλεκτρικέ παρατη... με για τις ηλεκτρικές μπαταρίες λόγω χάρη, το Όμπας λόγω χάρη που έχει έδρα στο ε, Μίσιγκαν. Ήδη έχει ένα μεγάλο κύκλο εργασιών, αλλά εάν προσελκυθούν και άλλες επενδύσεις θα υπάρξει αύξηση του δυναμικού. Εδώ λοιπόν οι διαπολιτιακές συμφωνίες ε, διευκολύνουν τα πράγματα. Έχουν περάσει αρκετέ δυνατότητε κατασκευή προ τι Ηνωμένε Πολιτείε και εδώ βλέπετε πάλι 50% στήριξη από τον δύο ή e στι Ηνωμένε Πολιτείε, 40% των παγκόσμιων κατασκευαστικών δυνατοτήτων ε, στι ηλεκτρικέ μπαταρίες ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε τεχνολογία του μέλλοντος. Αυτό που βλέπουμε στο μέλλον, μπαταρίε, υλικά, όλα αυτά επαναλαμβάνονται και σε άλλου τομεί, Τα προϊόντα βιοεθανόλη, λόγου χάρη, είμαστε πρώτοι στην παραγωγή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή στις δημοσιεύσεις. Αλλά βλέπετε πού πάει η κατασκευή. 5% έχουμε εμείς. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η κατασκευη 5 εχουμε εμει οι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Και όπου διαθέτουμε βασικά και σε καινούργιες εταιρείες, startups, πηγαίνουν στις ΗΠΑ. Παίρνουν δηλαδή τις καλύτερες εταιρείες μας, τις πιο ευθύς, γιατί εκεί έχουν καλύτερες συνθήκες για την κατασκευή. Η ίδια κατάσταση επαναλαμβάνεται σε πολλούς τομείς. Τα φωτοβολταϊκά λόγω χάρη, τελευταίο παράδειγμα, υπέροχο παράδειγμα για την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά. Εάν δεν μπορεί κανείς να πετύχει στη δική του την αγορά, τι να πω, εάν δεν υπάρχει πιο δυνατό μήνυμα, τι άλλο να πούμε. Στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχει εδώ μια εύρωστη αγορά, υπέροχη, στα διπλώματα ευρεσιτεχνία, στις δημοσιεύσεις, σε ό,τι αφορά την κατασκευή, σε όλη την αγορά συνολικά, παγκοσμίως έχουμε 13%. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν τα πάμε καλά. Όμως η ομάδα υψηλού επίπεδου έκανε μια μελέτη και σας δίνω εδώ τη σύνοψη. Μεταξύ του 2001 και του 2010 τι έγινε. Είχαμε έξι από τις κορυφαίες εταιρείες στα φωτοβολταϊκά έως το 2009 με μεγάλες πρωτοπολιέ των κυβερνήσεων, με μεγάλο μερίδιο της αγοράς, με την Επιτροπή να προωθεί την όλη αγορά. Το 2010 χάσαμε κάποια εταιρεία, την Q-Sales, και την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει καμία ευρωπαϊκή εταιρεία πλέον, ε, στις startups τουλάχιστον. Έχουμε χάσει την αγορά, έχουμε χάσει το μερίδιο μας την αγορά. Χάσαμε το δυναμικό μας να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παρ' όλα αυτά, από επιστημονική άποψη, είμαστε άριστοι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ επιθετικέ σε αυτόν τον τομέα. Δίνουν ε, επιδοτήσεις για την ε, ηλιακή ενέργεια, έχουν ειδικού νόμους Ανώνυμα μπορεί κανεί να κάνει έρευνα ή στην Ευρώπη δεν μπορεί, οπότε επιφυλάσσονται και οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Εν συντομία, αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι μια κοιλάδα του θανάτου. Έχουμε υπέροχη επιστημονική γνώση. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Επιστήμη χρηματοδοτεί κυρίω την επιστημονική έρευνα. Δυστυχώ όμω ξεχάσαμε πώς να χρηματοδοτήσουμε και πώς να περάσουμε από την αξία της επιστήμης ω την αγορά και τι θέσει εργασίας. Αυτό λοιπόν που αποφασίσαμε στην ομάδα υψηλού επίπεδου είναι να προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια γέφυρα ώστε να ενώσουμε τις δύο άκρες της Κοιλάδα του θανάτου. Έτσι φτάνουμε στις δράσεις καινοτομία και έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπαμε ότι έχουμε πολύ ωραία επιστημονική βάση και θέλουμε να την διατηρήσουμε αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε τα σανίδια ώστε να δημιουργηθεί η γέφυρα που θα μας οδηγήσει προς την αγορά. Πρέπει να μεταφραστεί λοιπόν η επιστημονική γνώση, να μετατραπεί σε τούβλα ε, γνώσης, τούβλα κατασκευαστικά για τον τομέα ακριβώς που μας απασχολεί προς την αγορά. Θα πρέπει αυτά τα τούβλα μετά να, να μετατραπούν σε πρωτότυπα προϊόντα και αυτό μέσα σε συγκεκριμένε γραμμέ, όπω αυτά που ακολούθησαν οι ΗΠΑ προκειμένου να προσελκύσουν εταιρείε. Μικρέ κινήσει, αλλά προσελκύουν μικρομεσαίε και ε, αφού φτιάξουν το πρωτότυπο, το ε, διαδίδουν στην αγορά και έτσι προχωρούν σιγά σιγά. Πρέπει λοιπόν τέτοια να προβλέψουμε. Παγκοσμίω ανταγωνιστικό κατασκευαστικό τομέα. Στον ε, κλάδο αυτό, από την επιστήμη στο προϊόν, Έχουμε το ε, τεχνολογική ετοιμότητα σε επίπεδο, όπω ονομάστηκε. Δεν θα σα δώσω πολλέ λεπτομέρειε για να μην βαρεθείτε, αλλά ω τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τη σοφία τη, ε, δημιούργησε μόνο τέσσερι πρωτοβουλίε. Εμεί ρωτήσαμε γιατί. Αλλά όσο περισσότερε ερωτήσει θέτουμε, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι, δεν υπάρχει, ότι υπάρχει κάποια προκατάληψη. Ιδεολογική, πραγματική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει να λάβει συγκεκριμένε συγκεκριμένα μέτρα για τη χρηματοδότηση των ΤΕΙ θα χρηματοδοτηθούν οι πρώτοι από, έως και την 8η μέχρι τώρα. Επίση, για περαιτέρω χρηματοδότηση σε αυτό το τομέα, θα πρέπει κάποια κονδύλια να μεταφερθούν για την ε, προώθηση τη ανάπτυξη των τεχνολογιών. Το υψηλό, το, η ομάδα υψηλού επίπεδου ε, έκανε κάποιε συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω χρησιμοποιώντα την βαθμονόμηση εδώ Πρέπει να είμαι πολύ απλό στην παρουσίαση δυστυχώ. Ε, το πράσινο είναι βασική έρευνα, το γαλάζιο η εφαρμοσμένη έρευνα και το χρώμα που επικρατεί, το κίτρινο, είναι η έρευνα ανάπτυξης κοντά στην ανταγωνιστικότητα. Βλέπετε τι κάνουν οι μεγάλοι μα ανταγωνιστές, η Κορέα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία. Στη βασική έρευνα έχουν όλοι επίπεδα κοντά στο 40%. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση 36% δαπανούν κατά όρο. Βλέπετε το σύνολο αυτό. Στοιχεία του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτά. Και μετά, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα, μα έχει πώ διαιρούνται όλα αυτά. Από 80 σε 92%. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε στο, στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής είναι ακριβώς το αντίθετο από πλευράς ε, θεμάτων έρευνας, το αντίθετο από αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ, Κορέα, Ιαπωνία κτλ. Ίσως είναι σωστό αυτό που κάνουμε και δεν χρειάζεται να αλλάξουμε, αλλά βρισκόμαστε στη μέση μιας ναι. μεγάλης κρίσης. Περιμένουμε λοιπόν να έχουμε μια έκθεση από τις ΗΠΑ αντίστοιχη με τη δική μας για τις κομβικές τεχνολογίες και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. 8 Ιανουαρίου δημοσίευσε μια έκθεση η αντίστοιχη υπηρεσία των ΗΠΑ για το πώς βλέπουν τη σύνθεση των θεμάτων ε, που θα χρηματοδοτήσει η δημόσια έρευνα και η ανάπτυξη. Εδώ βλέπετε ένα 24%. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μέσα σε μια κρίση πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα για τη βασική έρευνα ή όχι. Να τα στοιχεία ο νέος στόχος για τη βασική έρευνα είναι 17% και όχι 24% πια. Όλο και περισσότερο η εφαρμοσμένη έρευνα και η αναπτυξιακή έρευνα. Το ίδιο κάνει και η Κορέα, το ίδιο κάνει και η Σιγκαπούρη, από ό,τι ξέρω. Εμείς όμως είμαστε διαφορετικοί. Επειδή εστιάζουμε στη βασική έρευνα και στη βασική επιστήμη, στην Κομισιόν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας είναι μια συμμετοχή που μειώνεται στα προγράμματα έρευνα τη Κομισιόν. Αυτά είναι στοιχεία τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κόκκινο είναι το ποσοστό βιομηχανικών φορέων που συμμετέχουν, 39% στο 4 πρόγραμμα πλαίσιο, τώρα 25% στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα έχουμε ένα θαυμάσιο επιστημονικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρί συμμετοχή βιομηχανία, χωρί δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι σαφή όλα αυτά λοιπόν και πάλι η πηγή αυτών των στοιχείων είναι η ίδια η Κομισιόν. Οι συστάσει τώρα της Ομάδας υψηλού επίπεδου. Κάποιε από αυτές νομίζω θα σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική πολιτική βιομηχανία η οποία να οδηγείται από την ίδια τη βιομηχανία. Εμείς έχουμε αλληλεπιδράσει πολύ καλά με τις Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και υπάρχουν κάποιες συστάσεις που μπορείτε να κοιτάξετε και κάποιες από αυτές εμπίπτουν και στο δικό σας τομέα συζητήσεων στους επόμενους μήνες. Αυτές οι συστάσεις τώρα μπορείτε να τις συγκρίνετε και με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν μιλάει πια για να εκπαιδεύσει τον υπόλοιπο κόσμο λέει θέλουμε να φτιάξουμε νέες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους μας, τους πολίτες μας. Να ξαναέρθει η μεταποίηση, γιατί η μεταποίηση στη δημιουργία νέων προϊόντων είναι εκεί που δημιουργούνται νέα προϊόντα. Κοιτάξτε την ε, Apple που βασίζεται στις sketch, στις κύριες τεχνολογίες που δημιουργούν ικανότητες. Όταν δείτε λοιπόν αυτή την έκθεση, η πρώτη τους ε, πρόταση ήταν να αντιμετωπίσουν τα θέματα του, των τεχνολογιών, να επιταχύνουν τις διαδικασίες ε, ε, μεταποίησης με πιλωτικές γραμμές. Υπάρχει και το θέμα της μεταποίησης. Εμείς όμως δεν θα πρέπει να βάλουμε πιλωτικές γραμμές στα πανεπιστήμια, όπως λένε ορισμένοι, ούτε στους ερευνητικούς τομείς. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν στη βιομηχανία και μετά να προχωρήσουν οι ερευνητικοί φορείς να συνεργαστούν μαζί τους σε επίπεδο συμπληρωματικό. Και επίσης, αν δεν πιστεύετε εμάς, πιστέψτε τον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος ξέρει καλύτερα. Και έχει εμπειρογνώμα στα θέματα αυτά. Οι κέτς λοιπόν, οι τεχνολογίες αυτές, Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ακόμα μεμονωμένες, ε, απομονωμένες ε, διευθύνσεις γενικές που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, αλλά έχουμε και τις προκλήσεις για την κοινωνία. Και όπως άκουσα σε μια άλλη συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα αυτά είναι ασαφέστατα η πρόταση της Κομισιόν για το τι θα γίνει για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κοινωνίας είναι πάρα πολύ ασαφή. Μόνο μία πρόταση έχουμε που θα θέλαμε να ζητήσουμε από εσάς να υποστηρίξετε που είναι ότι όσο αντιμετωπίσουμε τις μεμονωμένες προκλήσεις της κοινωνίας θα χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς δομικούς λίθους για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αλλιώς αν υπάρξουν απαντήσεις που να χρησιμοποιούν εξωτερική τεχνολογία δεν θα έχουμε καμιά δυνατότητα να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να πιέσετε την Κομισιόν να υπάρξει μια πιο σαφής πρόταση από την Κομισιόν. Εν κατακλείδη. Πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση μας δίνει μια δυνατότητα να περάσουμε την κοιλάδα του θανάτου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι και να είναι βιώσιμη η χρηματοδότηση της έρευνας. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας που λέει 15 δισεκατομμύρια τη βασική έρευνα, μα δεν έχουμε τόσα χρήματα που να καλύπτουν τις βασικές αυτές τεχνολογίες από τις οποίες εξαρτάται όλη η βιομηχανία μας. Όλα αυτά φαίνονται και σε αυτά που δείξαμε. Είπαμε ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η πορεία. Υπάρχει μια γέφυρα που είναι πάνω από την κοιλάδα του θανάτου και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και σας ζητούμε να μεταλαμβαδεύσετε αυτό το μήνυμα στην Κομισιόν και να δείτε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Επειδή έχουμε, έχει περάσει ο χρόνος θα μείνουμε εδώ, δεν θα ανεβούμε στο Προεδρείο. Η κυρία Ρόιτοβα, η κυρία Ρούλα και ο κύριος Βάμπ θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Ξέρω ότι η κυρία Ρούλα και εγώ ενδιαφερόμαστε για κάτι που δεν το αναφέρατε, τις δημόσιες προμήθειες. Δεν το αναφέρατε λέω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της αμερικανικής επιτυχίας για το ξεπέρασμα της κοιλάδος του θανάτου. Παρακαλώ να το σχολιάσετε. Ρόιτο Βαρούλας Βάμπ. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμάσια παρουσίαση και τις ε, νέες κατευθύνσεις που προτείνετε σε σχέση με τα θέματα αυτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν, η οποία ήταν πολύ καλή. Είχα όμως ένα ερώτημα για τα θέματα αυτά. Λέτε ότι η καλύτερη παραγωγή και μεταφορά αγαθών θα πρέπει να έρχεται από τις χώρες όπου είναι πιο ε, φτηνή η παραγωγή. Οι φωτοβολταϊκές τεχνολογίες παραδείγματος χάρη. Αυτά είναι σημαντικά βιομηχανικά προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις η οποία θα εξασφαλίσει ότι εκμεταλλεύεται το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις τιμές. Και αυτό που θέλω να πω συνδέεται με το ερώτημα της κυρίας Ρόιτοβα. Δύο θέματα. Πρώτον, στη Γερμανία έχουμε την εμπειρία ότι στον των τομέων των φωτοβολταϊκών έχουν πάει όλα αυτά στην Κίνα, αλλά η βιομηχανία εργαλειομηχανών ουσιαστικά, των μηχανών που χρειάζονται για την παραγωγή φωτοβολταϊκών βρίσκονται στη Γερμανία και τα ηλεκτρονικά. Εγώ βρίσκομαι στη Βάδη Βιρτεβέργη από όπου προέρχεται η παραγωγή όλων αυτών των εργαλειομηχανών για τον τομέα αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Αν είναι τόσο φτι... φτηνές οι εργασιακές δυνάμεις σε άλλες χώρες, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το δικό μας δυναμικό που είναι η παραγωγή εργαλειομηχανών. Το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με την πολιτική που έχει ακολουθήσει η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια που έχει θέσει την έμφαση κυρίως στην παροχή υπηρεσιών. Αν αυτό είναι μια βιώσιμη αντιμετώπιση ή όχι. Και τέλος πιστεύω ότι τόσο στον τομέα των ε, κρατικών επιδοτήσεων και τη μεταρρύθμιση του θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περικόψουμε <clears throat> επιδοτήσεις που είναι νευραλικές για μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην μειώσουμε τη δική μας ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο, να μην περικόψουμε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι είναι καλό βήμα προς τα εμπρός οι καινοτόμες αυτές μορφές εταιρική σχέσης, αλλά η Κομισιόν αυτό το οποίο έχει προτείνει είναι ε, αυστηρές προδιαγραφές. Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς αυτές οι προδιαγραφές επιτρέπουν και τις καινοτόμες μορφές ε, ήταν ε, εξαιρετική η παρουσίαση. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ηλιακής ενέργειας που αναφέρατε. Ποιο είναι εδώ το θέμα κλειδί. Δεν συμφωνώ απολύτως με την κυρία Ρούλα ότι αν έχουμε τις εργαλειομηχανές τα έχουμε όλα. Υπάρχει και το θέμα της καινοτομίας και της δυνατότητάς της. Είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ηλιακή ενέργεια και τη χάσαμε. Δεύτερον, δεν θελήσατε να περιοριστείτε μόνο στη βασική έρευνα και επιστήμη, αλλά η Γερμανία και η Γαλλία πώς το βλέπουν. Και τέλος, είπατε ότι οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν πια τόσα πολλά δημόσια χρήματα, αλλά μήπως εννοείται ότι στην Ευρώπη είναι όλα πιο γραφειοκρατικά και πιο δύσκολα να διαχειριστεί κανείς. Τώρα εγώ. Το θέμα της εξάπλωσης των τεχνολογιών, όπως και εσείς είπατε, και οι πιλωτικέ δράσει, τα πιλωτικά προγράμματα είναι σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα. Ναι, είναι ζωτική σημασία. Το είπε η κυρία Ρούλε. Έχουμε το δυναμικό. Νομίζω το θέμα είναι η χρηματοδότηση. Εσεί είπατε ότι θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερα από τα κονδύλια τη έρευνα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια πραγματική πρόκληση αυτή. Να το σκεφτούμε τι μοντέλο έχουμε δημιουργήσει. Διότι είπατε κι εσείς ότι οι πολλές γενικές διευθύνσεις μοιράζονται την ίδια αρμοδιότητα. Αλλά θα έπρεπε να αναζητήσουμε και περισσότερα κρατικά κονδύλια. Μάλλον τα ιδιωτικά μπορεί να έρχονται από τη μία πλευρά, αλλά να συνδυάζονται με τα δικά μας στην κοινή χρηματοδότηση. Μόχλευση λοιπόν για περισσότερη ιδιωτική χρηματοδότηση. Εκεί μπορεί να είναι η απάντηση. Για το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει πρασίνισμα και στις τράπεζες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βοηθήσει και εδώ. Έχει γίνει μια επένδυση στον τομέα της έρευνας στην ανάπτυξη των πρώτων ιδεών. Αλλά δεν έρχεται χρήμα. Δεν τροφοδοτούνται όλα αυτά. Εκεί λοιπόν μια εταιρεία χρειάζεται να τροφοδοτηθεί. Δεν μπορεί να περιμένει δύο-τρία χρόνια για ένα εισόδημα. Αυτό είναι και η πραγματική κοιλάδα του θανάτου κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα τις απαντήσω με τη σειρά. Κυρία Ρόιτοβα, εδώ. Δεν μιλάμε για κατασκευή χαμηλού κόστους αυτή καθεύθυνση να σας δώσω μία περίπτωση για την ηλεκτρονική και μια, μια μονάδα ηλεκτρονικής. Μπορεί να είναι 5 δις ευρώ, μπορεί να είναι αυτοματοποιημένη μονάδα, αλλά δεν χάνουμε αυτού του είδους κομμάτια του κατασκευαστικού τομέα. Μιλάμε για ε, μονάδες συναρμολόγησης χαμηλού κόστους. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται ολοκλήρωση. Θα πρέπει να, συνεργα... να συνδυάζονται. Το καλύτερο παράδειγμα είναι να δούμε μια ευρωπαϊκή εταιρεία όπως η Nokia. Τι κάνει. Η, η αξία της Nokia χτυπήθηκε από το iPhone. Η μόνη εταιρεία που θα μπορούσε να απαντήσει σε μια τέτοια καινοτόμο κτέο του iPhone είναι η Samsung. Επειδή έχει αγοράσει την ηλεκτρονική και το λογισμικό, ώστε να φέρει στην αγορά πολύ γρήγορα ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν, είχαν μεταφερθεί ήδη εκτό Ευρώπη τα βασικά στοιχεία. Πρέπει κανεί να μπορεί λοιπόν, να συνδυάσει, να, να συναρμόσει τα διάφορα χαρακτηριστικά με διαφορετικού τρόπου, με υψηλή ποιότητα στοιχεία και εκεί μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εάν δείτε για το, τι γίνεται με το κόστος λόγου χάρη, 5 δις ευρώ, ε, το κόστος του μισθολογίου εδώ είναι πολύ χαμηλό. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είπατε επίση τα φωτοβολταϊκά. Ε, το αναφέρατε. Είναι ίση ώρα του παιχνιδιού εδώ. Σας έδειξα παραδείγματα των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν ένα, μια κρατική υπηρεσία το δικό τους ε, Υπουργείο ας πούμε, Ενέργειας για να απορροφούν τις δικές μας ε, εταιρείε και επιχειρήσεις με πρότυπα εγκαταστάσεων στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό δημιουργεί μερίδια στην αγορά, οπότε οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείε πάνε και αναλαμβάνουν δράση. Εκεί γίνονται μεγάλε επενδύσει. Όπω είπατε, το μεσαίο κομμάτι είναι το πλέον σημαντικό. Μπορούμε λοιπόν να του τυπήσουμε αν έχουμε ίσου όρου στο παιχνίδι. Φανταστείτε μια ευρωπαϊκή χώρα να προσπαθεί να προσφέρει πακέτα όπως των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι μόνο στους τομεί που ανέφερα, φωτοβολταϊκά, βιοεθανόλη. Δεν μπορούμε ακόμα να του ανταγωνιστούμε λόγω της νομοθεσίας μεταξύ άλλων. Η κυρία Ρούλε ανέφερε τα μηχανικά εργαλεία και τα μηχανήματα. Ναι, αλήθεια είναι. Η Γερμανία είναι, έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίω στα μηχανήματα, όμως τα τελευταία 10 χρόνια η Κίνα πέρασε στο 40% της παγκόσμιας αγοράς. Προχώρησε. Έχει ισχύοντα προγράμματα και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία με τις ακροάσεις που οργανώνουμε στο ομάδα υψηλού επίπεδου όπου απλώς αντιγράφει κάποια από τα βασικά μας ε, μηχανήματα και εργαλεία, όπως τα φωτοβολταϊκά. Η Κίνα έχει 40% λοιπόν της παγκόσμιας αγοράς για τα εργαλεία και τα μηχανήματα. Και εμείς δεν ακολουθούμε αυτήν την κατεύθυνση, παρόλο που η τάση υπάρχει και σε άλλους τομείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οι κατασκευαστές μηχανικών εργαλείων θα πρέπει να ετοιμάσουν τι επόμενες εκδοχέ, τις νέες γενιές των εργαλείων με συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής. Γιατί αν χάσουμε και την κατασκευή προηγμένου επίπεδου θα χάσουμε ήδη όλο αυτό το δυναμικό. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα στις, στους εξοπλισμούς λιθογραφίας. Υπάρχουν εταιρείε με πολύ καλή παραγωγή, αλλά δεν, αν δεν ετοιμαστεί εγκαίρως η επόμενη γενιά, εργαλείων θα χάσουν αυτό το δυναμικό. Η Γερμανία λοιπόν νομίζω κράτησε τη δυνατότητα της ε, καλής παραγωγής εργαλείων αλλά όχι το δυναμικό της κατασκευής. Τα μηχανήματα λόγου χάρη η Κίνα και οι Ηνωμένε θα αποβάλουν σε δοκιμίε πολύ γρήγορα και μετά τα βάζουν κατευθείαν στην αγορά. Είπατε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Νομίζω με τα προϊόντα που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές μας, ε, αλλού πρέπει να έχουμε το νου μας. Και προχωρώντας, το ανέφερε και ο κύριος Σφάμπ, τα φωτοβολταϊκά. Γιατί χάσαμε τόσο, πολύ, τόσο μεγάλο μερίδιο εδώ. Πρώτα απ' όλα γιατί η τεχνολογία για τα φωτοβολταϊκά δεν είναι τόσο προηγμένη τεχνολογικά όπως κάποιες τελευταίες εξελίξεις στην ανωτεχνολογία όπου πρέπει κανείς να δράσει γρήγορα. Στην παρουσίαση δεν είχα χρόνο να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αλλά θα βλέπατε ότι τα ποσά που διατίθενται για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας στην Κίνα ε, ξεπερνούν τις δικές μας δυνατότητες κατά πολύ. Ε, στην πραγματικότητα, ως τώρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ούτε καν αναγνωρίζει τη ΣΚΤΕ ως ξεχωριστή κατηγορία χρηματοδότησης. Και ένα σωρό ποσά πηγαίνουν στους τομείς αυτούς, αλλά είναι ένα μικρό κλάσμα, ένα μικρό τμήμα του τι συμβαίνει αλλού. Δεν ότι απλώς χρειάζομαστε περισσότερα χρήματα, πρέπει να δοθούν σωστές προτεραιότητες. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει και στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Κοινοτομίας. Όχι απλώς περισσότερα, αλλά σωστότερη θέση προτεραιοτήτων. Ο Φράνχοφ ήταν ε, μέλος της ομάδας υψηλού επίπεδου και σε κάποιους αυτούς τους τομείς ακολουθούσαμε το έργο που είχε προηγηθεί. Ο Φρανχόφερ λόγω χάρη στον τομέα τη ηλεκτρονική, είχε ήδη ετοιμάσει κάποια στοιχεία και ετοιμάσαμε ένα έγγραφο διαβούλευση. Το υποβάλαμε στην κυρία Κρούς, το υπέγραψε ο κύριος Φρανχόφερ και το είδανε ένα σωρό εταιρείε και πολλές γερμανικές Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε εδώ μια φωνή ενιαία, ένα ενιαίο μήνυμα από την Επιτροπή, αλλά ακόμα απομένει να δημιουργηθεί αυτό. Το τελευταίο σχόλιο ήταν από τον πρόεδρο της Επιτροπής σας, ότι το μεσαίο κομμάτι της γέφυρας είναι το πλέον καθοριστικό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα πρωτότυπα στην Ευρώπη. Ακόμη και αν μετά η μεγάλη συμβέλεια κατασκευή πάει αλλού. Εδώ πρέπει να παραδεχτώ ότι μας εξέπληξε ευχάριστα και αυτό που ετοίμασε η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών, οι οποίες μίλησαν για συνδυασμό χρηματοδότησης, όπως, όπως λέγω χάρη για ερευνητικό πρόγραμμα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Κοινοτομίας, με χρηματοδότηση τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών. Νομίζω στην ανακοίνωση για τις ΚΤΕ θα υπάρχουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Ελπίζω ότι σε αδρές γραμμές απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι. Νομίζω... Ναι, πρέπει να σας χειροκροτήσω μεν. Σας κατευχαριστώ γιατί κάνετε τον κόπο να προσέλθετε εδώ μέσα. Αφού χωνέψουμε την έκθεσή σας, θα δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. θα καταλάβατε κι εσείς ότι είμαστε, μας ενδιαφέρει πολύ η καινοτομία. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα των δημοσίων παρομήθειών, αλλά δεν θα γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα. Ελπίζουμε να παραμείνετε σε επαφή. Καλό είναι ότι αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου ε, γίνεται γνωστή. Θα θυμόμαστε το θέμα της κοιλάδας του θανάτου που μας είπατε. Και εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την φωτονική. Όλοι έχουμε κάποια σύνδεση στις περιφέρειές μας με πανεπιστήμια και άλλα μορφωτικά ιδουρήματα και θα συνεννοηθούμε και με τους εκπροσώπους των για να έχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ελπίζω να ξανάρθετε κάποτε να μας φωτίσετε ακόμη περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, εδώ λίγη η πρωινή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες. Θα ξαναβρεθούμε στις 3 για τις πολύ σημαντικές μας συζητήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουμε και ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ.